Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Η κυρία Ματσόνη θα φτάσει κάπως καθυστερημένα και θα έλθει εδώ στο Προεδρείο από τη στιγμή που θα φτάσει στην αίθουσα. Έχουμε το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης και αυτό είναι η οθέτηση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Να σας πω κάτι. Η συνάντηση των συντονιστών θα ξεκινήσει στις 11.30 σήμερα το πρωί και μετά θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα που την εβδομάδα που μας πέρασε έχει διανεμηθεί. Η κυρία Βίβιαν Reading, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έλθει εδώ και θα συμμετάχει στη συνάντηση το απόγευμα στις 4.30 και θα έχουμε τα στοιχεία, τα θέματα τότε με την ηθαγένεια και τα δικαιώματα των ε, πολιτών και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι επιβεβαίωσαν θα είναι εδώ από τους αναφέροντες θα είναι οι εξή. Στο σημείο 5 η 1335-208 σχετικά με την παραγωγή στο χρυσορυχείο του Τσελοπέκ στη Βουλγαρία και θα έχουμε εκπροσώπους από το ρηχείο που θα υποστηρίξουν την άποψή του στο σημείο 6. Η 1534 του 2008 για την αθλητικό τουριστικό κέντρο στην οριστερά της Ροδόπης και μετά η 1336-2008 σχετικά με την πλημελή λοπής δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία και μετά η 776 του 2009 σχετικά με τις παραβιάσεις χωροταξιών, χωροταξιών διατάξεων στο Χοντός Δος Φράιλες και το σημείο 10 το επόμενο σχετικά με Πολωνούς πολίτες που θέλουν ε, να ε, έχουν ε, του αυτού φίλου ζευγάρι. Και ακόμα έχει το σημείο 8 Εκεί θα ασχοληθούμε μετά από το 12. Πρώτα με το 12 και μετά με το 8 για τους κύριους και τις κύριες βουλευτές θα πούμε ότι θα έχουμε πιο πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκθεση του 2010 μετά από τη συζήτηση με την κυρία Ρέντινγκ. Το σημείο 2, ναι, καλημέρα, ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να σας πω τα εξής. Τη βδομάδα που μας πέρασε σας στείλαμε μια σημείωση σχετικά με την άνοιγμα και το κλείσιμο ορισμένων ε, αναφορών και ότι ε, θα, όσα ολοκληρωθούν θα συμπεριληφθούν ε, στα πρακτικά. Και δεν έχουμε στα διάφορα κάτι και μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εξέταση των αναφορών με το σημείο 4. Αλλά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ Το κύριο Μπουσούτιλ είναι απόν. Περιμένουμε λοιπόν, τον περιμένουμε και μεταξύ θα περάσουμε στο σημείο 5 που είναι για το περιβάλλον θέμα και έχουμε το πρώτο το 1335 του Χριστογένεφ βουλγαρικής ηθαγένειας συνοδευόμενη από 14.432 υπόγραφες σχετικά με την αύξηση της παραγωγής στο χρυσορυχείο του Τσελοπέχ στη Βουλγαρία. Ο αναφέρον είναι παρόν. Όχι, απόν επίσης. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ξεκινώντας. Ο κύριος Σιβανόφ έχει το λόγο. Βάσει των πληροφοριών που μας έδωσε ο αναφέρον, δεν μπόρεσε η Επιτροπή να δει ότι υπάρχει παραβίωση του σχετικού νόμου που αφορά αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η παραγωγή ξεκίνησε πριν από την προσχώρηση στην Βουλγαρία και η οδηγία για τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικές στην Βουλγαρία δεν εφαρμόζονταν τότε. Θα πρέπει να επιστρέψουμε προσοχή στο γεγονός ότι αυτό το επιχειρήμα αναφέρεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αξιολόγηση που άρχισε το 2004. Εάν υπάρχουν για το ίδιο θέμα ε, νέες ε, προτάσει θα εφαρμοστεί η διατάξη τη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι μετά από την ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 δεν έχει να προσέξει τίποτα. Ε, η Επιτροπή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στις 15 ε, Φεβρουαρίου 2010 η Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την ε, μελέτη την οποία είχε κάνει ο σχετικός Υπουργός Περιβάλλοντος σε σχέση με τα προβλήματα που αναφέρονται και την παραγωγή του χρυσορυχείου Τσελοπέκ. Σας ευχαριστούμε. Κάποιος που θα ήθελε να παρέμει πάνω σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε μία ερώτηση στην Επιτροπή για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε κάπως τα όσα ακούσαμε. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση κρατική, όπως έχει κατάσταση τώρα τουλάχιστον, επειδή είχε ενταχθεί η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την άδεια που δόθηκε για το πρόγραμμα αυτό αλλά στο τέλος σας είπατε γιατί το κονδύλιο έχει να κάνει με την ανεπάρκεια στοιχείων βάσει της οδηγίας Habitat. Στο 2010 η Εθνική Βουλγαρική Νομοθεσία είχε ακυρώσει τότε τις εκτιμήσεις επιπτώσεις του περιβάλλοντος σαν επαρκής εδώ τι γίνεται όμως. Έχουμε ένα πρόγραμμα που δεν έχει εκτιμήσεις. Άρα λοιπόν ε, είμαστε σε θέση σήμερα, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την εφαρμογή της οδηγίας Habitat για ενόψη μιας νέας εκτίμησης ε, που θα ρύθμιζε την κατάσταση. Ε, νομίζετε ότι η ανάλυση μου είναι η σωστή ή η κατάλληλη αυτή που κάνω τώρα. Ευχαριστώ. Ναι, στην Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κ. Μπουστινάρο. Θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με την ε, Μπελιέ, την διακεκριμένη συνάδελφο. Μετά από απόφαση του δικαστηρίου της Σόφιας, ότι στην αρχή της διαδικασίας δεν έγινε ΕΠΕ, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Πιστεύω ότι σήμερα η μόνη νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τη Βουλγαρία είναι η οδηγία Habitat και οτιδήποτε έχει σχέση με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος όπως και στις υπόλοιπες χώρες μέλη. Επισήμως, λοιπόν, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία και αν δεν εφαρμόζεται σωστά ή καθόλου η κοινοτική νομοθεσία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Διότι δεν μπορούμε να ζούμε ε, σε ένα κενό δικαίου για αυτή την περίπτωση στη Βουλγαρία, να δούμε ότι υπήρχε μία απόφαση πριν από την ε, πρόσβαση, ε, προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν χρειάζεται να γίνει τίποτε. Ακούστε είναι νομίζω ανάγκη οπωσδήποτε να ζητηθεί από τους επενδυτές και την βουλγαρική κυβέρνηση να κάνουν αυτή την ε, ΕΠΕ, δηλαδή την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ό,τι γίνεται να γίνεται τηρώντας την κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Εδώ Νομίζω ότι στο σημείο αυτό υπάρχει κενό έτσι όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς. Βέβαια, σχετικά με τα έργα, της επενδύσεις υπάρχουν πάντα ρυθμίσεις και ό,τι έγινε μετά από την ένταξη ενός κράτους μέλους. Νομοθεσία η οποία ενεκρίθη άλλωστε, μάλλον όσοι ίσχυε πριν από την ένταξη, τι να κάνουμε, αυτή είναι, αλλά μετά από την ένταξη θα πρέπει να είναι όλα αυτά σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Μετά από την ένταξη, επαναλαμβάνω, θα πρέπει κανείς να εξετάζει και να διαπιστώνει ποια είναι η επίπτωση των μέτρων αυτών που υιοθετήθηκαν όμως και πριν από την ένταξη και πώς επηρεάζουν τώρα πια το περιβάλλον και θα πρέπει κανείς να αναρωτηθεί, να πει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σχετικά έτσι και εδώ υπάρχει ένα κάποιο πρόβλημα γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει ρυθμισμένα. Κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται στη Βουλγαρία να υποβάλει το ερώτημα αυτό και να τους πει ότι πριν από την ένταξη αυτά τα και αυτά τα πράγματα και τώρα θα πρέπει να προβείτε σε μια μελέτη των μέτρων που υιοθετήσατε τότε. Έτσι, δεν τα αφισβητούμε αυτά που έχουν ληφθεί πριν από την ένταξη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τώρα των συνεπειών μια ανάλυση να γίνει και αυτή η εκτίμηση που προηγουμένη είπαμε δεν είναι δεσμευτική βέβαια, δεν είναι υποχρεωτική. Εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε μια μελέτη των επιπτώσεων αυτών των μέτρων από τη Βουλγαρία ή πρόκειται μόνο για μια εξέταση στοιχείων για όλα αυτά. Και τα κράτη-μέλη μερικές φορές μας λένε «Α, ό,τι κάναμε, κάναμε άλλο πριν από την ένταξη και άλλο το μετά την ένταξη γιατί ίσχυαν νομικά διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από την Επιτροπή αν είναι σε θέση δεσμευτικά, υποχρεωτικά να κάνει μια ανάλυση των επιπτώσεων και αν στέκουν τα πράγματα είναι σωστά έτσι νομικά. Ευχαριστώ. Just to make it brief, I we already... Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω το εξή. Όλες αυτές οι υποθέσεις τρελώνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δομίζω ότι δεν είναι ικανοποιητικό να έρχεται η Επιτροπή και να μας απαντά όπως απαντάει. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για να δούμε αν μπορούν να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των βουλγαρικών αρχών και της Επιτροπής για την περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο εκπρόσωπος επιτροπή έχει το λόγο και μετά θα υποβάλω και εγώ μια πρόταση. you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Officer Brickland. Πρώτα απ' όλα, για την νομοθεσία που αφορά τις περιβαλλοντικές ε, επιπτώσεις. Εάν πριν από την προσχώρηση είχε γίνει είχε δοθεί η άδεια, ισχύει άλλη νομοθεσία και αν μετά η κοινοτική νομοθεσία. Δεδομένου τώρα ότι πρόκειται για νομοθεσία σε θέματα δικασίας την εφαρμόζουμε μετά και όχι πριν συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, αν είμαστε από του Natura 2000, έτσι όπως είπε η Σαντρίν Μπελιέ, θα μπορούσαμε ακόμη να έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Βεβαίως δεν μπορείτε να κάνετε αναδρομικά την ε, μελέτη επιπτώσεων, αλλά έχετε στα πλαίσια της Natura 2000 την υποχρέωση να ελεγχιστοποιήσετε τους κινδύνους. Εδώ όμως δεν πρόκειται για χώρο ο οποίος καλύπτεται από την ε, Natura 2000, άρα δεν εφαρμόζεται εδώ η οδηγία ε, Habitat. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχετε μία επιστολή από τον ανάδοχο του σχεδίου που λέγει ότι ο επενδυτής εγκατέλειψε το έργο αυτό, πράγμα το οποίο βάζει τέλος σε αυτό το θέμα. Δεν θα γίνει τίποτε σε αυτή την περιοχή λοιπόν. Βεβαίως αν είσαστε στην ε, κάτω από την οδηγία Natura 2000 θα γίνονταν περαιτέρω μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν έχουμε όμως αυτή την ε, περίπτωση τώρα, δεδομένου ότι όπως σας προανέφερα ο επενδυτής εγκατέλειψε την ιδέα. Ήρθε ο αναφέρον κύριος Γκαμπρινόφ πριν να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό, θα του δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα λάβω το λόγο εξ ονόματος όλων των συναδέλφων που έχουν καθαθέσει μία αναφορά για αυτό το θέμα του χρυσορυχείου του Τσέλοπεκ που χρησιμοποιεί μία τεχνολογία θέλησε να χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία την οποία τελικά εγκατέλειψαν. Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχουν και μία σειρά μη κυβερνητικών οργανώσεων που προσέφυγε στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Βουλγαρίας το οποίο αποφάσισε ότι η μελέτη για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είχε γίνει σωστά, δεδομένου ότι δεν είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανόνες και κάποια θέματα που αφορούσαν διαβούλευση των κατοίκων της περιοχής. Έτσι λοιπόν προς το παρόν εγκαταλείφθηκαν αυτά τα σχέδια σε δύο άλλες περιοχές κοντά σε μια στο Ετσολή και σε μια μικρή πόλη κοντά στο Λοβτίβ αναφέρουν κάποιοι ότι χρησιμοποιείται η ίδια τεχνολογία με αυτή που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν καταρχάς και στο ξεροχείο του Τσέλοπεκ, δηλαδή τη μέθοδο έκπληξης με κιανούχες ενώσεις. Το θέμα είναι η δημόσια διαβούλευση. Κοντά στο Πλόβδιβ η διαβούλευση έλαβε χώρα μόνο σε ένα μικρό χωριό, το Κλόκλαν, στο οποίο ζουν περίπου 7.000 άτομα και στο Plovdiv είναι 10 χιλιόμετρα πιο μακριά και εκεί ζουν 300.000 άτομα. Η διαβούλευση όμως έγινε μόνο στο μικρό χωριό των 7.000 κατοίκων. Έτσι, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι δεν ζητήθηκε η άποψη των πολιτών όπως θα έπρεπε από τους ενδιαφερόμενους. Αυτό λοιπόν έκαναν οι βουλγαρικές αρχές. Πάρθηκαν λοιπόν κάποιες αποφάσεις χωρίς να ληφθεί υπόψη η θέση που θα εξέφραζαν όλοι οι κάτοικοι, οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της περιοχής αν είχαν ερωτηθεί. Εμείς στο Πλόβδιβ μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε 14.000 υπογραφές κατά της χρησιμοποίησης αυτής της μεθόδου, δηλαδή την έκπληση με κιανούχος ουσίες και θα θέλαμε να απαγορεύσετε τη χρησιμοποίηση αυτή της μεθόδου έκπληση με κιανούχες ουσίες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στη Βουλγαρία όπως και στη Ρουμανία οι δυνατότητες που έχουν οι κυβερνήσεις μας και η διαφθορά θέτουν σε κίνδυνο την ε, δημόσια υγεία. Αυτά θέλαμε να πούμε στα πλαίσια αυτής της ε, αναφοράς. Ο κύριος Μπουστινάρο. Δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα, υποστηρίζω αυτά τα οποία είπε ο Αναφέρον. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια πραγματική λύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι με μεγάλη, πολύ μεγάλη ψηλοψηφία ζητήσαμε όλες οι διαδικασίες που αφορούν τα χρυσορυχεία να μην χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους των καινούχων ουσιών. Δεύτερον, με αυτή την περίπτωση της Βουλγαρίας το Τσέλοπέκτς, Έχουμε μία ειδική περίπτωση. Κατά κάποιο τρόπο μία νομολογία, όπου οι νόμοι που εφαρμόστηκαν στην περίοδο πριν από την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχαν σύμφωνα με το δικαστήριο στη Σόφη. Και δεύτερον, τουλάχιστον θεωρητικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν ζήτησε στον επενδυτή τον Βούλγαρο να εφαρμόσει σωστά την μελέτη αυτή για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ό,τι έγινε πριν από την ε, ε προσχώρηση έχει καλός, αλλά οτιδήποτε γίνεται μετά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα επιπτώσεις της μελέτης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή η περίπτωση μπορεί να είναι παρεμφερείς με άλλες που συμβαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε την επίσημη ερμηνεία όλων των παρομοίων περιπτώσεων από την Επιτροπή. Δηλαδή, εάν οι νόμοι που εφαρμόστηκαν πριν από την προσχώρηση εφαρμόστηκαν σωστά και μέχρι πότε. Σήμερα όμως ο μόνος νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί είναι αυτό της μελέτης για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και αν, βλέπετε στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν σώθηκε η κατάσταση μετά από την ε, τρομερή ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά διότι ο επενδυτής ε, απέσυρε το ενδιαφέρον του. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Δεν θα πρέπει οι επενδυτές, ε, οι ανάδοχοι έργων να βασίζονται σε προενταξιακές νομοθεσίες για να κάνουν ό,τι θέλουν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει στηθεί αρκετά ήδη. Τελευταίο και μετά εγώ θα υποβάλω μια πρόταση. Ναι, και εγώ μία πρόταση, δεν ξέρω τι γίνεται αν καταλήξαμε όπως πρέπει, αλλά ιδιαίτερα αρνητικά τα διατυπώνουμε τα πράγματα εδώ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όταν μία χώρα έχει κάτι το αρνητικό σαν νομοθεσία στο το περιβάλλον, να χορηγεί άδειε και μετά να γίνεται μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά λέει Α, ακούστε αυτό που έγινε πριν, δεν μα ενδιαφέρει και πολύ εδώ τώρα. Όχι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε που δεν είναι αυτό. θα πρέπει να διεξάγεται ένας διάλογος με τα νέα κράτη-μέλη και με τα νέα κράτη-μέλη γενικά. Όταν ακριβώς ε, να πρέπει να δούμε πώς ρυθμίζουμε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και να τα εξετάζει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος για να έχουμε και περαιτέρω συντονισμό γιατί από τη στιγμή που κάνουμε χρήση μιας υπάρχουσας τεχνολογίας θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς με ποιο τρόπο θα εφαρμόζονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε συνεχώς να λέμε «Α, αυτό είναι παλιά, αυτό είναι καινούριο» και η Επιτροπή να λέει «Εμείς δεν έχουμε παραπερισμένη ε, νομική αρμοδιότητα σχετικά με αυτά επειδή πρόκειται για θέματα παλιά και ότι παρόλο που υπάρχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εντάξει, με τους, ε, σχετικά με την γεωργία, ε, μπορούμε, ίσως κάναμε με τον αρμόδιο οργανισμό, ρυθμίσαμε τα πράγματα, αλλά για το περιβάλλον πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η αναχθολογία και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έχουμε διαπιστώσει. Ότι ε, είπαμε ότι επιθυμούμε να απαγορεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι και η κυρία Μπελιά και οι υπόλοιποι έβαλαν το, θέσαν το θέμα όπως πρέπει. Θα πρέπει στην Επιτροπή να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει πληροφορίες σχετικές από το κρατομέλος, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και νομίζω ότι η τελευταία αυτή ε, ε, το τελευταίο αίτημα είναι σωστό να πάει ταυτόχρονα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό για μια γνωμοδότηση. Θα πρέπει να παραμείνει αυτό το θέμα και να μας προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες και αυτό το τι γινόταν πριν από την ένταξη και μετά την ένταξη θα πρέπει το θέμα αυτό να λυθεί στα πλαίσια των ε, ευρωπαϊκών οδηγιών και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα παιδιτικοί με οποιασδήποτε δραστηριότητε ε, σημειώνονται από τη χώρα. Και ε, θα περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 6 Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα επιστρέψουμε στο πρώτο σημείο, το 4. Ο κ. Μπουσούτιλ θα θέλαμε να τον καλωσορίσουμε και να δώσουμε το λόγο για το σημείο 4. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να ερωτήσω αν είναι εδώ αναφέρον για να μπορέσει να λάβει το λόγο. Δεν είναι εδώ αναφέρον από ό,τι κατάλαβα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα αρχίζοντας να υπενθυμίσω στα μέλη περί τίνος πρόκειται, δηλαδή να μιλήσω για την οδηγία σχετικά με τι παραπληκτικέ πρακτικέ των εταιρεών έκδοση καταλόγων επιχειρήσεων. Πολλέ φορέ τέτοιου είδου επιχειρήσει προσεγγίζουν ΜΜΕ και διάφορες οργανώσεις καθώς και επαγγελματίες και ατομικά κάποια άτομα του στέλνουν μία αίτηση στην οποία καλείστε να εγγραφείτε ε, δωρεάν σε μία εταιρεία έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων. Και αφού εγγραφείτε, παίρνετε ένα λογαριασμό για χίλια ευρώ το μήνα και το ότι δεσμεύεστε για τρία χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι παραπλανηκτικό κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει παντού στην Ευρώπη και πολλές ΜΜΕ και πολλές ελληνικές οργανώσεις, σχολεία και δημόσιες βιβλιοθήκες είναι ε, θύματα αυτής της παραπλάνησης. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συμβαίνει ε, και σε επίπεδο διασυνοριακό. Δηλαδή, κάποια επιχείρηση είναι ε, εγκατεστημένη σε μια χώρα και μια επιχείρηση που τέτοιου είδους βρίσκεται σε μια άλλη χώρα και την παραπλανά. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Γι' αυτό ε, έχουμε σήμερα αυτή την έκθεση εδώ. Πρέπει να πούμε ότι πολλές δεκάδες τέτοιου είδους αναφορές έχουν υποβληθεί. Το Δεκέμβριο του 2009 εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε μία έκθεση ψήφισμα την οποία εκπώνησα εγώ και ζητούμε από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ενεργήσουν ώστε να βρουν μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Ιδιαιτέρως κάναμε στην έκθεση αυτή τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπογραμμίσαμε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα, διότι όλο περισσότερα άτομα γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, τόσο λιγότερα θα παραπλανηθούν. Επίσης, ζητήσαμε να υπάρχουν λύσεις διαμερθωριακές για το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για τέτοιου είδους θέμα. Επίσης, τρίτη παρατήρηση, ζητήσαμε να εφαρμόζεται περισσότερο η κείμενη νομοθεσία κοινοτική, διότι δεν νομίζω ότι εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία την κοινοτική τα κράτη-μέλη. Τελικά ζητήσαμε από την Επιτροπή να αλλάξει την νομοθεσία εάν δεν είναι επαρκώς ε, σωστή, αποδοτική και αποτελεσματική αυτή η νομοθεσία κοινοτική. Δυστυχώ, παρά αυτή την σαφή διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραμένει το πρόβλημα και επιτρέψτε μου να πω ότι κατά κάποιο τρόμα το πρόβλημα πρέπει να πω ότι ακόμη χειροτέρεψε, διότι Τώρα πρόκειται για πραγματική βιομηχανία. Δεν πρόκειται απλώς ε, για μία απάτη που κάνει μία επιχείρηση, αλλά για μία βιομηχανία απάτης που δημιουργεί πολλά προβλήματα και ζημιώνει τις επιχειρήσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Για να ε, αναφέρω κάποια παραδείγματα. Η έκθεσή μου βασίστηκε σε αναφορά κατά της European City Guide, με έδρα την Ισπανία, ε, από την ε, Βαρκελόνη πήγε στη Βαλένσια, η έδρα αυτής της επιχείρησης, αλλά και σε άλλες ε, χώρες, η Construct Data στην Αυστρία, Νόβα Τσένια στην Ελβετία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με την οποία έχουμε στενούς εμπορικούς δεσμούς και άλλες εταιρείες EU Business Services, Expo Guide, DAT και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Τι προτείνω λοιπόν εγώ κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο προτείνω είναι ως Επιτροπή το θέμα, να ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα αυτό και να επιμείνουμε μέχρι να μας αποδείξει η Επιτροπή ότι πραγματικά μπορεί να βρει μια πραγματική λύση, δεδομένου ότι πάρα πολλά άτομα ακόμη είναι θύματα αυτής της απάτης. Πολλά άτομα κάθε μέρα λαμβάνουν πληθώρα επιστολών νομικού περιεχομένου και απειλητικών από αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτά θέλω να πω. Ελπίζω ότι θα έχω την υποστήριξη των συναδέλφων και θα ήθελα να υποβάλουμε μία προφορική ερώτηση, ερώτηση στην Ολομέλεια, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε στην Ολομέλεια το θέμα αυτό με παρουσία της Επιτροπής, αλλά να παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη των πραγμάτων μετά από την προφορική ερώτηση, να κάνουμε και μια έκθεση, να ψήφισμα και να ζητήσουμε να διευθετηθεί το θέμα αυτό το οποίο χρονίζει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μποσούτιλ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπη Επιτροπή, τον κύριο Βιέκο. Ευχαριστώ. Γνωρίζει βεβαίω η Επιτροπή τις απάτες αυτές και κυρίως αυτές των directory companies και ότι και όντως αυτές οι επιχειρήσεις προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε έναν αριθμό επιχειρήσεων μικρών και μεσαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη και άλλων επαγγελματιών. Τώρα, εξακολουθεί να λαμβάνει παράπονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις απαντήσεις της η Επιτροπή λέει ότι όντως υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τέτοιες πρακτικές, κυρίως παραπλανητική διαφήμιση, ότι ισχύει η νομοθεσία αυτή και στις χώρες μέλη και ότι από όσα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις επαφές με τις χώρες μέλη, οι εθνικές αρχές παρακολουθούν και ασκούν διώξεις όσο μπορούν καλύτερα. Η Επιτροπή συνέχισε φέτος να ενθαρρύνει τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ε, προβαίνουν στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η οδηγία. Το οποίο μας φέρνει στα θέματα που θέτει ο αξιότιμος ε, βουλευτής κύριος Μπουσουτήλ στο ψήφισμά του του Δεκεμβρίου του 2008 και στο πλαίσιο αυτό σημείωσε η Επιτροπή, σημείωνε μάλλον στην απάντησή της τότε, ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις σπανίως άγουν τα θύματά τους ενώπιον των δικαστηρίων, διότι είναι απολύτως απίθανο οποιοδήποτε δικαστήριο να κρίνει υπέρ των επιχειρήσεων αυτών. Ταυτόχρονα η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα επιβολής της νομοθεσίας λόγω του διεθνούς χαρακτήρα των απατών αυτών. Τόνιζε ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν οι πρακτικές αυτές είναι να ε, αυξηθεί η γνώση περί των απατών αυτών μέσα στην επιχειρηματική κοινότητα. Και μέσα στο 2009 συνέχισε να παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ιστοσελίδες και άλλους ιστοτόπους και διεπίστωσε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται πολύ εντονότερα σε διάφορες ε, ιστοσελίδες επιχειρήσεων που ασκούν τις απάτες αυτές και σε επιχειρήσεις και σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων που φαίνεται ότι έχουν γνώση πλέον του ενδεχόμενου του κινδύνου απάτης. Βέβαια, το πρόβλημα παραμένει. Και το νέο στοιχείο τώρα απέναντι στην παλαιότερη απάντηση της Επιτροπής προ τον κύριο Μπουσουτήλη είναι ότι η Επιτροπή η Κομισιόν δηλαδή αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ανάληψη νομοθετική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό και ιδίω την έγκριση ανακοίνωση για τις ε, απάτες αυτές που θα ε, εκδοθεί περί τα τέλη του 2011 και στην βάση της ανάλυσης των επιχειρήσεων αυτών θα προτείνουμε και σε ποιους τομείς μπορεί να αναθεωρηθεί η οικία οδηγία. Θα ξεκινήσει μια μεγάλη διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμμετοχή και των χωρών μελών και άλλων ενδιαφέρομενων μερών ε, των οργανώσεων εκπροσώπησης επιχειρήσεων των διαφόρων δικτύων Enterprise Europe Network και άλλα για να διεξαγάγει αυτή τη διαβούλευση. Στα πλαίσια του εγχειρήματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει όλες τις πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες για να ανακοπεί αυτή η δραστηριότητα και όπως σημειώνει η Επιτροπή στην απάντησή της τον κύριο Μπουσουτήλ θα εξετάσει αν είναι σωστό να μπουν ειδικέ διατάξεις στην και οδηγία για να αποτρέπονται τέτοιου είδους πρακτικές διατάξεις παρόμοιες με αυτές που περιλαμβάνονται σε άλλες οδηγίες. Επίσης, θα εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να επεκταθούν τα όργανα της νομοθεσίας που έχουν σχέση με την επιβολή της νομοθεσίας αυτής στην οδηγία περί ε, καταπολέμησης απατηλής διαφήμισης μπορούν, μπορεί να περιληφθούν και νέες διατάξεις που να ενισχύουν την διαμεθοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών. Βέβαια, μια τελική, μια τελική ε, λύση για να βελτιωθούν οι κανόνες κατά της απατηλής διαφήμισης θα εξαρτηθεί και από τα πορίσματα της ε, δημόσιας διαβούλευσης την οποία αρχίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Τσίτσεστερ ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σάιμον Μπούσουτιλ για τη δουλειά που έκανε στον τομέα αυτό και που έχει ικανοποιήσει πολλούς από τους ψηφοφόρους μου, διότι πολλοί μου έχουν γράψει παραπονούμενοι για τις απάτες αυτές και, για τις, και εξηγώντας τις προσωπικές τους εμπειρίες, τους απάντησα στέλνοντα αντίγραφο της εκθέσεώς του, ε, μαζί και με ορισμένες συστάσεις των δικών μας τοπικών ε, αρχών που είναι αρμόδιες για ε, το, τις εμπορικές επιχειρήσεις στην χώρα μου υποστηρίζω την ανάγκη να αναλυφθεί δράση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, διότι είναι διεθνές το θέμα, όπως εξήγησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεφεύγουν σαν χέλια οι άνθρωποι αυτοί, στέλνουν απειλητικές επιστολές, εκφοβιστικές επιστολές στους ε, παραλήπτες και πρόκειται για μια αποκρουστική πρακτική η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει. Στη δική μου περίπτωση ένας αριθμός ψηφοφόρων μου μου έχουν γράψει. Φαίνεται να υπάρχει μια νέα παραλλαγή σε αυτή την ε, συνηθισμένη απάτη, την οποία εξηγούν στις επιστολές τους και έχω γράψει επίσης και έχω ε, πληροφορήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω να υπάρχουν κάπου οι επιστολές μου στα αρχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνουν παραδείγματα αυτών των απατηλών πρακτικών. Και χαίρομαι που η Κομισιόν σχεδιάζει αναθεώρηση τη οδηγία. Υποστηρίζω τον κύριο Μποσουτήλ, πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και πρέπει με τον τρόπο αυτό να προσπαθήσουμε να καθησυχάσουμε και τους ψηφοφόρους μας που έχουν πέσει θύματα παρόμοιων απατών. Το καλύτερο, συμφωνώ και εγώ, είναι η σωστή ενημέρωση, η πληροφόρηση. Έχω εκδώσει ανακοινοθέντα τύπου στον τοπικό τύπο της εκλογικής μου περιφέρειας, αλλά είναι λιγάκι σταγόν εν το ωκεανό, διότι ως γνωρίζετε ο τύπος δεν ασχολείται ιδιαίτερα με ανακοινοθέντα τύπου, δυστυχώς των Ευρωβουλευτών, δυστυχώς λέω. Παρ' όλα αυτά ας κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ λοιπόν και εσάς κύριε Πρόεδρε και εσάς Σάιμον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 Muchas gracias, señor Yar. Κυρία Χέφνερ, κυρία Ματίθαρ, άλλο. Κάτι ήθελα να πει καινούριο ο κύριο Χέφνερ. Συγγνώμη. Δύο σύντομε ερωτήσει, αν επιτρέπετε. Όποιο υφίσταται τέτοια πίεση μπορεί να αντιδράσει με βάση το αστικό δίκαιο και συνήθως στα γερμανικά δικαστήρια τουλάχιστον τον ε, δικαιώνουν. Εδώ όμως με ενδιαφέρει και η ποινική διάσταση. Αν μπορεί δηλαδή να περιγραφεί στον νόμο ως ποινικά διοκόμενο αδίκημα, ώστε να διώκεται αυτεπαγγέλτος, αντί να είναι υποχρεωμένος κάθε φορά ο, ε, στη ζημία να προσφεύγει στα αστικά δικαστήρια. Και για την οδηγία τώρα προστασίας των καταναλωτών μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις της, ώστε ε, βασιζόμενοι σε αυτές να ψηφίσουμε μια πιο ξεκάθαρη ε, ρύθμιση. Ο κ. Μποστινάρου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αρκετές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να χαιρετήσω την όλη πρωτοβουλία και το θάρρος που επέδειξε ο κύριος Μπουσούτιλ. Όλα αυτά δείχνουν καθαρά ότι η Επιτροπή μας, ναι, μπορεί να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, ακόμα και όταν ε, τα κράτη και οι διάφορες επιτροπές ε, δείχνουν την αδυναμία τους. Το πρόβλημα, τα πρόβλημα έχει οπωσδήποτε να κάνει με κάτι που είχε να κάνει με το πέρασμα του χρόνου και κάθε φορά το τι γινόταν. Μας μίλησαν για ό,τι γινόταν και οι εθνικές διατάξεις για να αντιμετωπιστούν παρόμοιες απάτες φαίνονται ότι είναι ανεπαρκείς, τουλάχιστον, τουλάχιστον. Βέβαια, οι νομοθετικές ευρωπαϊκές πράξεις, οι δικές μας και αυτές δεν επαρκούν, σίγουρα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά νομικά κενά, τα οποία τελικά είναι υπέρ των ε, ανθρώπων αυτών με τις παράνομες ενεργές τους. Πολύ συχνά ε, τα θύματα σε ένα κράτος ε, δεν μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη απέναντι σε μια εταιρεία που εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την έδρα της. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αποζημιωθεί το θύμα απάτης. Είναι σαφή και συγκεκριμένα τα πράγματα λοιπόν. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να εκφράσω την υποστήριξή μου στον κύριο Μπουζούτιλ και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτεχύνει όλη διαδικασία και την εκτίμηση σχετικά με την ανάγκη νέων νομοθετικών πράξεων, νέων εργαλείων. Θα ήθελα να ζητήσω και από τα κράτη-μέλη να πάρουν πραγματικά ιδιαίτερα στα σοβαρά τις συστάσει του κύριου Μπουσούτιλ και να μα ενημερώσουν εμά εδώ στην Επιτροπή για όλε αυτέ τι συζητήσει, για όλα αυτά

τα πραγματικά τεράστια σημασία θέματα και τολμάω να ελπίσω ότι το θέμα αυτό που είναι πραγματικά εύκολο για να λυθεί να ε, ε, αποδειχτεί κιόλα ότι η Επιτροπή είναι ε, υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ των πολιτών και νομίζω ότι έτσι θα δείξουμε καθαρά ένα τομέα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα περίπλοκο, απλά και μόνο να δείξουμε το βαθμό αποτελεσματικότητα ε, στα όργανα Ευχαριστούμε. Ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Ρίκο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέθηκαν διάφορες ερωτήσεις εάν το ουσιαστικό δίκαιο εφαρμόζεται ορθά, εάν η νομοθεσία είναι επαρκής. Ζητήσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει γρήγορα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και με κατάλληλη νομοθεσία. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει καλά την οικονομική ζημία που επιφέρουν οι απάτες αυτές τις μικρές επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά την ενόχληση και σε ό,τι αφορά την οικονομική ζημία. Το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το διαμεθοριακό. Συχνά οι επιχειρήσεις που ασκούν τις απάτες έχουν την έδρα τους εκτός των ε, περιφερειών δικαιοδοσίας όπου είναι, των δικαστηρίων δηλαδή όπου είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις που αποτελούν τα θύματα. Υπάρχουν παραδείγματα βέβαια συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά δεν είναι επαρκή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα το ουσιώδες δίκαιο, υπάρχει η σχετική νομοθεσία και με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις προετών ένα τσεχικό δικαστήριο ε, παρέκλεινε από την ε, συνήθι, συνήθως ασκούμενη πρακτική. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει πώς μπορεί να κάνει σαφέστερη την νομοθεσία, ώστε να δείχνει πιο ξεκάθαρα ότι είναι απαγορευμένες οι πρακτικές αυτές. Από την άλλη μεριά, είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα, και εκεί θα πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερα το βάρος των προσπαθειών μας, να εξεύρουμε τρόπο δηλαδή να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Όπως γίνεται και στον χώρο προστασίας των καταναλωτών, ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ζητούν δικαστική και άλλη αρμόδια αρρωγή από τις ομόλογες αρχές τους στις άλλες χώρες μέλη. για να διωχθεί η επιχείρηση που ασκεί την απάτη. Μιλώντας για την οδηγία προστασίας καταναλωτών, μία από τις επιλογές που ανέφερα πριν είναι ο νόμος που απαγορεύει τις αθέμητες πρακτικές και περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις ήδη, τις οποίες θα μπορούσαμε είτε να αντιγράψουμε ή τουλάχιστον να τις θεωρήσουμε ως πηγή εμπνεύσεως για να επιλέξουμε άλλες ορθές ε, νομοθετικές διέταξεις. Ωστόσο, διαβεβαιώνω τα αξιότιμα μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό. Αρχίζουμε τώρα δημόσια διαβούλευση και διαδικασία αναθεωρήσεως, νομοθετική δηλαδή, που θα οδηγήσει μάλλον σε αναθεώρηση της οδηγίας κατά της απατηλής διαφήμισης, που θα αλλάξει ήδη τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, είτε θα εξοπλίσει την ε, οδηγία αυτή με κάποιες προβλέψεις για ενισχυμένη δικαστική συνεργασία. Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ πρώτα όλους και όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν για να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία μου. Πρωτοβουλία που είναι πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως πρωτοβουλία υπέρ όλων των θυμάτων που μας έχουν ε, υποβάλει τα παραπονά τους. Ακόμα και ευρωβουλευτές έχουν λάβει τέτοια έντυπα. Είναι ξεδιάντροποι αυτοί οι απατεώνες επιχειρηματίες. Δεν θα πω οι ευρωβουλευτές την πάτησαν τελικά, ας το πούν οι ίδιοι αν θέλουν. Αλλά πρόκειται πραγματικά για έσχος και χρειάζεται να σταματήσει αυτό. Χαίρομαι πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει και νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος όταν ακούω την Επιτροπή να λέει ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 2011, για να δούμε την πρωτοβουλία αυτή. Σήμερα είναι μόλις η 1η Φεβρουαρίου. Μέχρι το τέλος του έτου σημαίνει στην ουσία άλλον ένα χρόνο. Άρα θα προσθεθούν χιλιάδες ακόμη θύματα. Άρα θα παρακαλέσω, θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί ταχύτερα. Δεν είναι, κάποιο, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο φάνηκε τώρα για πρώτη φορά. Εδώ και χρόνια παραπονούνται και μας καταγγέλουν οι πολίτες ε, τις απάτες αυτές. Επίσης, προσοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να αλλάξουμε το δίκαιο. Σε άλλες περιπτώσεις λέει έχουμε ήδη το δίκαιο, είναι, υπάρχει ήδη το δίκαιο. Α αποφασίσει τέλο πάντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν έχουμε τις απαραίτητες νομικέ διατάξεις, τότε έχει το καθήκον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ώστε οι χώρες μέλη να εφαρμόζουν, να επιβάλλουν τις διατάξεις αυτές. Εάν όχι, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, αν δεν το πράξουν αυτό οι χώρε μέλη, τότε πρέπει να ε, ξεκινήσει διαδικασίε σε παραβάση. Δεν υπάρχουν όμω τέτοιε, εάν από την άλλη μεριά το εφιστάμενο δίκαιο δεν είναι επαρκές, τότε χρειάζεται να αλλάξει ώστε να γραφτεί στις μαύρες λίστες η πρακτική αυτή άπαξ και διαπαντός. Και ένα τελικό σχόλιο. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά αποτρεπτική λύση. Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να πέφτουν θύματα και να έρχονται σε εμά να ζητούν βοήθεια. Δεν θέλουμε να γίνουν θύματα. Καν. Ποτέ. Αυτό είναι που επιθυμούμε και γι' αυτό χρειάζεται να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να κοπεί από την ρίζα της αυτή η απατηλή διαφήμιση. Προτείνω λοιπόν να υποβάλουμε προφορική ερώτηση, αστεθεί αυτό υπόψη των συντονιστών, προφορική ερώτηση με ψήφισμα που να εξασφαλιστεί η συνέχειά του μετά με δραστηριότητες της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Θα ήθελα εκ μέρου όλη τη Επιτροπή να σας ευχαριστήσω για το επίπεδο των απαιτήσεών σας. Θα πρέπει όντω να είμαστε πολύ απαιτητικοί ώστε τέτοιου είδου απάτε προς ΜΜΕ να μπορούν να τύχουν άμεση ανταπόκριση από την Κομισιόν. Να μην περιμένουμε. Νομίζω ότι σωστά εσείς ε, ε παρουσιάσατε αυτές τις απαιτήσει στο κατάλληλο επίπεδο. Και όπως λέτε σωστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την παρούσα νομοθεσία να θέσει σε εκείνη όλους τους μηχανισμούς ε, παραβίασης και να μην καθυστερήσει μέχρι το τέλος του χρόνου πριν να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απέτηση στην οποία θα πρέπει να διαβιβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι όπως είπατε κυρία Μπουσούτιλ θα πρέπει με την κείμενη νομοθεσία να αρχίσει να επιβάλλει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και να μην περιμένει την νομοθετική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει όντως να είμαστε απαιτητικοί. Βεβαίως Πιστεύω ότι η πρότασή σας να γίνει στην Ολομέλεια προφορική ερώτηση με ψήφισμα θα πρέπει να προχωρήσει και θα αποτελέσει και ένα καθαρό μήνυμα προς τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί αυτό το μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είμαστε να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε αυτού του είδους τις απάτες. Συμφωνούμε λοιπόν με την ιδέα σας και σας ευχαριστούμε γιατί βάλατε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Περνούμε στο επόμενο θέμα. Σημείο 6. Αναφορά Βορισλάβ Σαντόφ, βουλγαρική Ιθαγέννη, ξενόμαστε εταιρείε αγροτικών και περιβαλλοντικών έργων. Νομίζω ότι έχουμε μαζί μα κάποιο εκπρόσωπο των ε, αναφερόντων. Ε, θα ήθελα να σα πω ότι έχουμε καθυστερήσει πολύ. Παρακαλώ λοιπόν και τον αναφέροντα και του συναδέλφου να είναι πάρα πολύ σύντομη για να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλα τα σημεία της σημερινή διάταξης. Ο αναφέρον παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να παρουσιάσω κάποια γεγονότα η οροσυρά της Ευρώπης, της Ροδόπης, είναι πάρα πολύ σημαντική στα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά. Και η υψηλότερη οροσυρά είναι στα 2.000 μέτρα. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομορφιάς περιοχή που προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και τέσσερα χρόνια και η υποχρέωση των αρχών μας είναι να προστατεύσουν από την καταστροφή όλες τις περιοχές που ε, καλύπτονται από την Νατούρα ε, με από παράνομες, παράνομα κτίσματα και καταστροφή. Ε, προβλέπεται να γίνουν κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις στο τουριστικό κέντρο Πέρελικ εδώ βλέπετε τον υπεύθυνο του έργου. Έχει πρόκειται για μια offshore εταιρεία με έδρα την Κύπρο που θέλει να κτίσει. Υπάρχει μεγάλα σχέδια για να χτιστούν εγκαταστάσεις σκι και ξενοδοχεία σε δυναμικότητα σχηλίων κλινών στην περιοχή. Σταμάτησε το σχέδιο αυτό κάποια στιγμή αλλά σήμερα για την αναφορά αυτή έχουμε μια απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο τμήμα της πρότασης για το αθλητικό και τουριστικό κέντρο στο Περελίκ πήρε άδεια, προετοιμάζεται τελή κατασκευή. Αυτό όμως δεν είναι αληθές, διότι η εταιρεία αυτή έκτισε στην ε, κορυφή της οροσυρά, στο Πέρελικ, αυτό το κτίσμα. Αυτό είναι το κτίσμα λοιπόν. Είναι παράνομο και σε αυτή την περιοχή η εταιρεία έχει βάλει αυτές τις πινακίδες που είναι παράνομες Κάναμε έκκληση εθνικές αρχές για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. και να αποκαταστήσουν την περιοχή και να γκρεμίσουν αυτό το παράνομο κτίσμα και, θέλουμε, και έχουμε υπογραφές για να υποστηρίξουμε αυτή την αναφορά εκ μέρους όλων των κατοίκων, διότι δεν πρέπει να καταστραφεί αυτός ο οικότοπος που προστατεύεται από την Natura 2000, το δίκτυο. Εκ μέρους της Επιτροπής ο κύριος Ιβάνοφ. With regard to petition 1534 of 2008, the Commission services have έχουν ενημερωθεί οι, επιχειρή... οι αρχές υπηρεσίες της, Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατασκευή του τουριστικού και αθλητικού κέντρου χωρίς πρώτα περιβαλλοντική μελέτη σύμφωνα με την οικία οδηγία της 92.43 η, εφαρμογή, η υλοποίηση του έργου θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στο οικολογικό περιβάλλον της Ροδόπης και ιδίως της κορυφής Πέριδικ. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγαγαν έρευνα και έθεσαν το θέμα υπόψη των βουλγαρικών αρχών που οδήγησε σε τροποποίηση της ε, οικίας νομοθεσίας που έλαβε και έλαβε απόφαση το Κοινοτικό Συμβούλιο της περιοχής του Μαρτίου 2009. Τροποποίηση δηλαδή του χωροτακτικού σχεδίου, που δεν έγινε όμως ποτέ τόπου δεν έγινε πραγματικά επί του εδάφους. Στο φως των μέτρων που έχουν λάβει οι βουλγαρικές αρχές, και παρόλο που το Γενικό Χωροτακτικό Σχέδιο εγκρίθηκε, δεν εφαρμόστηκε. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις μελλοντικέ εξελίξεις σε σχέση με το Αθλητικό Κέντρο Περιλίκ και θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από τον αναφερόμενο σχετικά με το θέμα αυτό. Θα του διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε από τις βουλγαρικές αρχές και βρισκόμαστε σε τακτική επαφή μαζί τους για να ε, παραμείνει θετική η κατάσταση. Κύριε Άουκεν. Ευχαριστώ. Θα τονίσω την ανάγκη να διεξαχθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή στη Βουλγαρία. Τίθενται πολλά θέματα εδώ. Ασφαλώς και θα πρέπει να μπορεί να γίνει στα πλαίσια επίσκεψη αυροφροσύνη. Πάντοτε θα πρέπει να είμαστε ευγενεί, πάρα πολύ ευγενεί, αυροί. Αλλά όχι όμως επίσκεψη αυροφροσύνη. Θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες, τι οικονομικές δυνατότητες που μας δίνει το επίδομά μας. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται κάποια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από πλευρά τη Ευρωβουλή για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Μποστινάρου. Πρόεδρε, να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Άουκεν. Θα είμαστε ευγενείς, αλλά δεσμευμένοι, στρατευμένοι όμως, διότι εδώ βλέπουμε να παίζεται ένα παιχνίδι πραγματικά εξαιρετικά περιορισμένης εφαρμογής των διατάξεων. Μετά το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την μη ορθή υλοποίηση του χωροτακτικού σχεδίου που ενέκρινε το Κοινοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αρκείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιες επίσημες πληροφορίες που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή, αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο, καμία ένδειξη, εάν εφαρμόζεται το σχέδιο ή όχι και η ίδια ύπαρξη του κτηρίου αυτού που βλέπουμε στην φωτογραφία και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, δεν ζήτησε καν ποτέ να κατεδαφιστεί το κτίριο και να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Πρόκειται για πλήρη παράληψη εφαρμογής των υφιστάμενων δικαιικών κανόνων. Άρα συμφωνώ απολύτως με την ε, αποστολή εξεταστική των πραγμάτων επιτροπής επιτόπου και βεβαίω να είμαστε όχι μόνο ευγενεί, αλλά να πάμε να ψάξουμε ακριβώς τι γίνεται εάν υπάρχουν παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων και εν τέλει πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιόν μας με ξεκάθαρες πληροφορίες, γιατί αυτές οι ασαφείς πληροφορίες που μας δίνει δεν είναι μόνο άσχετες, είναι απολύτως απαράδεκτες. Έρχεται εδώ η Επιτροπή και μας λέει «Α, βασιζόμαστε πληροφορίες που μας δίνουν οι αρμόδιες ε, τοπικές αρχές που έχουν μεν εγκρίνει αλλά δεν εφαρμόζουν κτλ». Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Ποστινάρο και κύριε Βιντιέρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Προς την αυτή κατεύθυνση με όσους πήραν τον λόγο προηγούμενα. Είναι τρία τα θέματα. Το πρώτο όμως που δείχνει ότι δεν γίνεται σεβαστή η ρύθμιση Natura 2000 για τη βιοπικιλότητα στην ε, ε, Βουλγαρία και εκεί είναι από τα θέματα που θα ασχοληθούμε που πρόκειται για το ποια θα είναι αυτά τα σημεία της Natura 2000 και αυτά στη Βουλγαρία. Όχι μόνο σε αυτά που έχουν οριστεί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία αλλά δεν ξέρουμε και τι γίνεται με ποια θα οριστούν σε παρόμοια σημεία. 20 χρόνια περίπου μετά από το κείμενο για την οδηγία του 92 Habitat και εν ώψη της νέας στρατηγικής βιοπικιλότητας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους μήνε θα μας υποβάλει θα ισχύει για τα δέκα επόμενα χρόνια για τα νέα κράτη που εισήλθαν, εντάχθηκαν και για τη Βουλγαρία. Η κατάσταση εκεί θα πρέπει να μας απασχολεί, να μας ενδιαφέρει και υποστηρίζω την πρόταση μιας επιτόπου επίσκεψης και έρευνας και ακόμα περισσότερο αυτά να γίνουν τάχιστα Είμαι υπέρ του η Επιτροπή Αναφόρας να έρθει σε επαφή με τις κυβερνητικές βουλγαρικές αρχές, να τις προσκαλέσουμε να έρθουν εδώ στο Ευρωπαϊκό να μας πούν πως έχει κατάσταση για την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τη βιοπικιλότητα και μάλιστα στο χώρο ακριβώς, το βουλγαρικό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε ο Η κυρία Γκουτιέρες έχει το λόγο. Δεν ήθελα κανονικά πρώτο λόγο, αλλά κάτι ήθελα να πω ότι τελικά πέρασα όλη μου τη ζωή δίνοντας μάχη για να ε, τα προστατεύσουμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, ε, εδώ το πρόβλημα είναι ότι σαν πολίτες, ε, οι πολίτες θέλουν να υπερασπιστούν το χώρο αυτό με ένα μόνο όργανο εργαλείο που είναι το Natura 2000, ενώ πρόκειται για επιτόπου αρχές που είναι αρμόδιες ή κρατικές. Και εδώ έχουμε αυτούς καταλόγους από όλα αυτά τα προβλήματα ότι παραβιάζουν αυτούς τους χώρους, τους φυσικούς, λόγω κακό διαχείρισης του ε, εκεί από τις τοπικές αρχές ε, μαζί και με τις δημοτικές αρχές. Και εδώ λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε ακριβώς κοντά στον πολίτη, ότι αν ε, υπάρχουν αλλού αρμοδιότητες, εκφορούνται αρμοδιότητες, τότε βλέπουμε τη διαφθορά. Και πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα όπως πρέπει αλλά εδώ έχουμε τα εξή ε, τέσσερα άτομα που απασχολούνται ας πούμε εκεί. Και εδώ ίσως αποτελεί μια ητοπία το να δώσουμε τη μάχη γιατί δεν είναι μόνο το πράγμα με το Natura 2000, είναι ο χώρος ο φυσικός όλα αυτά και μόνο με τους ε, τομείς αρμοδιότητας κατάλληλους εκεί μπορούμε κάπως να πετύχουμε γιατί ε, ε, το Natura 2000 ε, το παρακάμπτουν τα κράτη-μέλη και δεν μπορούμε έτσι να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κουτιέρες, λέει και ο Πρόεδρος. Βέρμαν. Ja, danke schön. Ich möchte mich auch den Kollegen anschließen, die meinen, dass eine fact finding Mission hier mehr als angebracht ist. Νομίζω ότι το ερώτημα πρέπει να τεθεί πώς είναι δυνατόν να χτιστεί σε μια κορυφή βουνού ένα τέτοιο κτίσμα χωρίς να το πάρουν χωρίς να ε, ασχοληθεί κανείς. Πράγματι, μια επίσκεψη επιτόπου είναι πραγματικά σημαντική και θα έπρεπε όλοι να εμφανιστούμε με μια ενιαία φωνή. Ασφαλώς ευγενής, ασφαλώς ωστόσο αποφασισμένη, αλλά κάποια στιγμή και η ευγένεια πάβει όταν παραβιάζεται ξεκάθαρα ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Γιάρα. Συμφωνώ απολύτως με όλους τους προλαλήσαντες. Μία ερώτηση, συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το μέγα αυτό ε, έργο, στα σχέδια δηλαδή, έχει, τα σχέδια έχουν αποσυρθεί. Το κτίριο αυτό εντάσσεται μέσα στο μεγάλο αυτό έργο. Το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απεσύρθη ή δεν απεσύρθη το σχέδιο. Η κυρία Γιώτοβα. Ακούστε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πρόταση των συναδέλφων για εξεταστική επιτροπή στην Βουλγαρία. Δεν είναι και η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε παραβιάσεις των διατάξεων του Natura 2000 στη Βουλγαρία. Και ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη. Προδιετίας αρχίσαμε να εξετάζουμε τα προβλήματα των πουλιών και των ε, οικοτόπων τους, των βιοτόπων τους. Ε, καμία από τις συστάσεις, σας βεβαιώνω, που ακούστηκαν εδώ, που έκανε δηλαδή η Επιτροπή Αναφορών, καμία από από τις συστάσεις που έκανε είτε η Επιτροπή Αναφορών είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόστηκαν. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι συζητούμε, στέλνουμε κάποιους στη χώρα μέλος, κανείς όμως τελικά εκεί δεν θεωρεί ότι έχει την ευθύνη να εφαρμόσει τα όσα προτείνουμε. Διερωτώμε λοιπόν και πάλι οι συζητήσεις που κάνουμε. Ο κόσμος που έρχεται εδώ να παρουσιάσει τις αναφορές του, τι νόημα έχει. Και ιδίω όταν γνωρίζουμε τα προβλήματα επιτόπου, το γεγονός ότι η κοινοτική αρχή δεν έλαβε απόφαση ή η απόφαση ελήφθη αλλά ε, δόθηκε η έγκριση αλλά μετά ήρθε η έγκριση, θα ξαναδοθεί η έγκριση. Σας βεβαιώνω ότι στην διετία που θα ακολουθήσει το κτίριο που βλέπετε εκεί στην κορυφή δεν θα μείνει μόνο του, δεν θα είναι το μοναδικό. Όπως και για τις ανεμογεννήτριες στην Βία Μπάντικα, έρχονται και μας λένε «Άμα δεν μπορούμε τώρα να κατεδαφίσουμε πράγματα που ήδη έχουν χτιστεί». Συμφωνώ λοιπόν με εκείνους που λένε ότι χρειάζεται νέα επίσκεψη στη Βουλγαρία και είναι καιρό πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει και μια σύνοψη για τα ποια πράγματα, με ποιες συστάσεις τελικά συμμορφώθηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, ορίζουμε μία ζώνη στο δίκτυο Natura 2000 και τι κάνουμε μετά. Στο θέμα του ορισμού έχει αρκετά υψηλό ποσοστό η Βουλγαρία. 7% είναι οι κακοί μαθητές, η Μεγάλη Βρετανία 8 η Δανία, ο μέσος όρος ο κοινοτικός 15, η Βουλγαρία 34%. Και βεβαίως, εάν κρυστεί ένα σπίτι στη μέση μια τόσο μεγάλης εκτάσεως, δεν φαίνεται αμέσως. Τι είναι σημαντικό, ο έλεγχος. Έχουμε τόσους πολύ μεγάλους ε, οικοτόπους που ανήκουν ε, στο Natura 2000 που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους και πρόκειται για 26.000 τέτοιους οικοτόπους και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να εκλεγούν. Για την ε, προστασία λοιπόν όλων αυτών των οικοτόπων του δικτύου 2000 έχουμε πρόβλημα δεδομένων. Εμπιστευόμεθα του αναφέροντο, τον κύριο Τζαντόφ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα κάνουμε επίσκεψη τόπου τον Απρίλιο. Βεβαίω είμαστε υπέρ όλων των πληροφοριών, τι οποίε θα μπορούσαμε να έχουμε από τη δική σα επιτροπή. Έχουμε την έκθεση επίσκεψη που έγινε στη Βουλγαρία του 2008. Πρόκειται πρωταρχική σημασία πληροφορία για μα. Όλο περισσότερε πληροφορίε λοιπόν έχουμε για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μα, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε του κανόνε. Στο ερώτημα του κύριου Γιάρ, τώρα θα απαντήσω ότι εφόσον απεσύρθη το εν λόγω σχέδιο, μάλλον πρόκειται για κάτι το οποίο είναι παράνομο και για το νομοθεσία της Βουλγαρίας. Αλλά βεβαίως θα ζητήσουμε επαλήθευση της κατάστασης επιτόπου από τις βουλγαρικές αρχές, όπως θα το κάνετε και εσείς όταν πάτε επιτόπου, όπως και εμείς. Ακούσαμε όλες τις ε, απόψεις και νομίζω ότι η άποψη πληροψηφία είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι παραμένει εκρεμής η αναφορά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους τις προφορίες που μας έστειλαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες προφορίες μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια αυτής της αναφοράς θα ζητήσουμε περισσότερες προφορίες από τις βουλγαρικές αρχές και εγκρίνουμε επισήμως την επίσκεψη μίας αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας επί τόπου, συνεντεύξεις ε, με μέλη από τη διοίκηση, με τους αναφέρτους, για να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια σε όλες αυτές τις αναφορές που αφορούν το θέμα αυτό και την προστασία του περιβάλλοντος. Το επόμενο θέμα που θα εξετάσουμε επίσης, θα το συμπεριλάβουμε στην επίσκεψή μας. Περνούμε στο σημείο 7, τελευταίο σε σχέση με τη Βουλγαρία. Και δεδομένου ότι είπαμε ότι θα πάμε στη Βουλγαρία, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Ο κύριος Κόβατσεφ, αναφέρω να έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής σας αφορούν και την επόμενη περίπτωση, την επόμενη αναφορά και πάλι έχουμε μία περιοχή κοντά στα παράλια του Ευξήνου Πόντου που καταστράφηκε. Εδώ βλέπετε τον ποταμό Βάια που καταστράφη το 2007, εξαφανίστηκε ο ποταμός και οι βουλγαρικές αρχές στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτησαν υπάρχει αποκατάσταση. Αλλά το καλοκαίρι του 2009 βλέπετε στη διαφάνεια ότι δεν έγινε τίποτε για την αποκατάσταση του ποταμού. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να γίνουν τα πράγματα όπως στο παρελθόν, να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Στην αναφορά αυτή, σε σχέση με την Natura 2000, στην Οροσιρά Ρίλα έγινε μία αναφορά για την ε, προστασία της αρκούδας. Ξέρουμε ότι είπαν ότι θα πρέπει η περιοχή αυτή στα Ρίλα να θεωρηθεί ως προστατευμένη ζώνη. Επίσης, Όταν θα κάνετε την επίσκεψή σας επί τόπου θα σας δοθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες και αιτιολογημένε. Πολύ καλά. Θεωρώ ότι ε, ολοκληρώθηκε εκεί η συζήτηση αυτού του θέματος, δεδομένου ότι στην επίσκεψη ε, θα συμπεριληφθεί και αυτό το μέρος που αναφέρεται εδώ στην αναφορά αυτή. Λοιπόν, είπαμε ότι το 8 θα το συζητήσουμε μετά το 12. Περνούμε λοιπόν συζήτηση του σημείου 9. Αριθμός 1098 παρουσίαση από τον Χουαν Αντώνιο Καράσκο Ράχελ. Εξ του φορέα Πλαταφόρμα Πορελεστούδιο Επιδημιολόγικο για την εκπόνηση ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη για του κατοίκου τόσο τη Κομιτεία του Γιβλαρτάρ όσο και του Γιβλαρτάρ. Από την Επιτροπή ο κ. Βάχτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με αυτή την αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι ήρθε σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές και άρχισε έρευνα για την εφαρμογή της ε, οδηγίας της σχετικής οδηγίας. Σήμερα τα, απο, τα πορίσματα που διαθέτουμε δείχνουν ότι υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις της εγκατάστασης αυτής, αλλά γίνονται διορθωτικές δράσεις. η επιχείρηση που ε, ασκεί τη λειτουργία της ε, εγκατάστασης ήδη επενδύει και σχεδιάζει και μελλοντικά επενδύσεις για την βελτίωση των τεχνικών ώστε να μειωθεί ή να αρθεί απολύτως η ε, ρήπανση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της αρμόδιας αρχής και αυτές έχουν περιληφθεί στην σχετική άδεια, στην σχετική έγκριση ε, λειτουργίας. Βασισμένη στα γεγονότα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Κάποια παρέμβαση μήπως, κάποιος που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Θα θέλαμε εδώ να έπρεπε να κάνει τις 26 Απριλίου έπρεπε να είχε συζητηθεί πέρυσι και θα πρέπει να γίνει μια επιδημιολογική έρευνα για τους κατοίκους εκεί στο Γιβραλτάρ και όσο γίνεται καλύτερα συμπερισμένα και στείλαμε μια επιστολή και στις δύο αρχές για την ε, μελέτη αυτή, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία απάντηση από πλευρά τους. Άρα ε, λοιπόν παραμένει ανοιχτή η αναφορά αυτή, ε, περιμένοντας, αναμένοντας την απάντηση από τις αρχές. Και τώρα πάμε στο σημείο 10 του κυρίου Μπέρν Χόφμαν γερμανικής ηθαγένεια, σχετικά με την ε, εικαζόμενη εγκαστική αγορά και κατάχρηση κοινωτικής χρηματοδότησης στο Έλτσε, επαρχία του Αλικάντε. Ο κ. Βλότς από την Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο αναφέρον μιλά για εικαζόμενη αναγκαστική αγορά και κατάχρηση κοινοτικής χρηματοδότησης στο ΕΛΤΣΕ. Και αναφέρεται επίσης ε, σε ανεπαρκή υποδομή σχετικά με το δίκτυο υδροδότης και ηλεκτροδότηση και το αποχευτικό δίκαιο. Αναφέρεται σε διάφορους ισχυρισμούς που είχε απευθύνει χωριστά και στην Όλαφ, Όσον αφορά την ε, χωροταξική διάταξη που προβλέπει οι, προβλέπουν οι τοπικές αρχές, θέλουμε να πούμε ότι αυτά τα θέματα είναι περιφερειακής εθνικής νομοθεσίας και δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τα μη επαρκή έργα υποδομής στον τομέα της ίδρευσης και της επεξεργασίας λιμάτων. Αναφέρουμε τη σχετική οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και για την προστασία των ε, υδάτων το Μάιο του 2010 αποφάσισε η Επιτροπή να ε, προσφύγει στο δικαστήριο κατά της Ισπανίας για ε, λυπή ε, για μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της οδηγίας και η γνωμοδότηση του δικαστηρίου ήταν κατά της Ισπανίας διότι δεν εφαρμόζει τις κατάλληλες ε, διαδικασίες για την διαχείριση και την προστασία των υδάτων. Πρέπει επίσης να πω ότι κάποια από τα επιχειρήματα του αναφέροντος δεν καλύπτονται από την κοινοτική αρμοδιότητα. Το θέμα επίσης των ε, καταχρήσεων που αναφέρονται έχουν εξεταστεί από εμάς για θέματα προστασίας των υδάτων. Έχουμε ασχοληθεί, θα ζητήσουμε την Ισπανία να έχει την καλά τάλληλη υποδομή για να μην υπάρχει πρόβλημα με τα θέματα της προστίας των υδάτων και υδροδότης αυτής της περιοχής του Σέλτσε, όπως αναφέρει ο Ευχαριστώ, κύριε Άουκεν. Πρέπει να σας πω ότι με απογοητεύει πάρα πολύ η Επιτροπή όταν λέει ότι δεν υπάρχει θέμα παρέμβαση επιτροπή. Όταν παρουσίασα την έκθεση, εγώ είχα, με ζητήσει με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή να κάνει κάτι, να παρέμβει. Είπαμε ότι επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει και προσφυγή στα μέσα για τέτοιου θέματα. Το ίδιο είχε γίνει και για τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, για άλλες χώρες. Αυτά έλεγε η έκθεση. Και τώρα που έχει ψηφιστεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια το ανέφερε. Το θεωρούσε και ως σημείο αναφορά η Κομισιό. Και ζητήσαμε από την Επιτροπή να λάβει το θέμα αυτό πολύ σοβαρά υπόψη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που συνεχίζεται. Δεν έχω τις τελευταίε προφορές στη διαθέσή μου, αλλά πόσον γνωρίζω και κρίνω, τέτοιου είδους παραβιάσεις βασικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε μία ιδιοκτησία παραβιάζονται. Τώρα μας λέει η Κρός Επιτροπής ότι είναι θέμα εθνικής δικαιοδοσίας και απευθυνθείτε σε αυτούς. Όσον αφορά το θέμα του ύδατος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το θέμα της προστασίας των υδάτων, αλλά βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι δεν προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους και μιλούμε για πολίτες, όχι μεγάλες επιχειρήσεις. Παρακαλώ λοιπόν να παραμείνει ε, η υπόθεση αυτή, να μην κλείσει. Θέλει κανένας άλλος συνέλφος το λόγο. Άρα λοιπόν Παραμένει ανοιχτή η αναφορά αυτή και θα δούμε την κατάσταση σχετικά με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, όπως είπε η κυρία Άουκεν άλλωστε. Το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι το 11 και ο αναφέρον είναι παρόν. Είναι ο κύριος Γκόρντον Μπέλ του κ. Ρόλαν Σάρπ, Βρετανική Ιθαγένεια, εξ ονόματο της Εθιωθών Ντεβεθίνο Ντεοντών, Χέντελο Φράιλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ πολλού άλλου πολίτε ε, που ζουν στην περιοχή μου στην ε, Ισπανία και εκπροσωπώ τουλάχιστον 500 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζοντας, θα πω ότι πιστεύουμε τους στόχους και τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία που μας προσφέρει η κοινοτική νομοθεσία. Όλοι έχουν το δικαίωμα να κατέχουν ε, περιουσιακά στοιχεία, να έχουν μία ιδιοκτησία και όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει την δέσμευση να προστατεύουν τα βασικά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών όταν γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο σημαντικό όμως θέμα είναι η προστασία της ζωής μας και μετά της ιδιοκτησίας μας. Αλλά η ζωή μας, εάν δεν προστατεύεται, η ιδιοκτησία μας έχει μεγάλη σημασία. 16 χώρες 16 χρόνια μετά την προσχώρηση της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την απέτηση να αισθανόμαστε ασφαλείς στις, ε, στα σπίτια μας. Το 2005 θεσπίστηκαν ε, νέες ε, πολεδομικές δραστηριότητες στα πλαίσια της οικοινής ε, ανάπτυξης της ε, ε, περιοχής μας. Είπε, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η υπεύθυνη ότι στα ε, χωριά μας, στο Χοντόντες Λας Νιέβες, προβλέπονται σύμφωνα με τα νέα οικιστικά ε, σχέδια να κτιστούν 10.000 νέα σπίτια, τουλάχιστον για 25.000 περισσότερους ανθρώπους. Ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα με την υδροδότηση της ε, ε περιοχής. η οποία δεν έχει ε, Παρκή είδωτα και βεβαίως μάθαμε ότι τα οικιστικά σχέδια στην, ε, σύμφωνα με τον Ισπανικό νόμο επιτρέπουν στην ε, κυβέρνηση να υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες να δώσουν το 40% της γης την οποία κατέχουν και να πληρώνουν και 60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ώστε να διατηρήσουν την υπόλοιπη που έχουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί απειλή για 60 ιδιοκτήτες σπιτιών στην περιοχή μας. Το οικιστικό και στεγαστικό σχέδιο στους Φράιλες και στο Χοντόλ Νιέβες λέμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επίσης προβλέπεται όταν χτιστούν, ε, χτιστεί αυτός ο νέος οικισμός ότι θα υπάρξουν ε, σχέδια για την διάνοιξη δρόμων. Αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία συμβαίνουν επανειλημμένως και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στην Ισπανία. Ε, η Επιτροπή σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την εν λόγω κατάσταση δεδομένου ότι έχουν γίνει και διάφορες επισκέψεις ερευνητικές και στην Ισπανία και ε, η κυρία Άουκεν έχει κάνει μία πρόσφατη επίσκεψη στην οποία ζήτησε να σταματήσει η κοινοτική χρηματοδότηση προς την Ισπανία εάν δεν εφαρμόζει σωστά την κοινοτική νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει όταν μια ευρωπαϊκή χώρα, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερο από 25 χρόνια, με την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εποφελείται θετικά από την ε, κοινοτική χρηματοδότηση και, και συνεχίζει να εφαρμόζει ε, νόμους και πρακτικές που είναι εντελώς αντίθετης προς την ε, δεύτερο πιο σημαντικό θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών υπάρχει ε, πρόβλημα. Σας ευχαριστώ κύριος Ράμος εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μην τα συνοψίσω όλα αυτά γιατί ο αναφέρον ε, ήδη μας ε, έκανε την περίληψή του σχετικά με όσα έχουν γίνει σχετικά με αυτό και θα θέλω να συμπληρώσω ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν την αναφορά αυτή σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινοτικό δίκαιο το οποίο είναι εφαρμοστέο εδώ σε θέματα περιβάλλοντος. Η χωροταξική οργάνωση εδώ στο Φράιλες, στο Αλικάντε κοντά στη Βαλένθια και ακριβώς η χωροταξία του περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών όπως και το δικαίωμα δικαιοσύνη και το αναγκαστική απομάκρυση σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, το κρατικό, το εθνικό και όχι το κοινοτικό τώρα εδώ στην όλη χορταξικό σχεδιασμό. Αυτό που θα πρέπει βέβαια να γίνει σεβαστό είναι το δίκαιο το κοινοτικό που θα πρέπει να εφαρμοστεί εδώ. Ε, έχουν σημασία οι οδηγίες σχετικά με τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικές ε, στρατηγικής σημασίας, ε, σχετικά με σχέδια και προγράμματα, όπως επίσης και φυσικού χώρου σχετικά με τα πτηνά στο Habitat και εδώ στο το χωροταξικό αυτό σχέδιο για να έχει επηρεάσει τα πράγματα, ακριβώ όταν παίζει τα πράγματα στο Natura 2000 και το για το Ίδωρο, η 2060, η οδηγία και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαχείριση, κατάλληλη διαχείριση και διάθεση των ε, πόρων ύδατο στην περιοχή. Και εδώ, σύμφωνα με αυτό το φάκελο, χρειάζεται, βλέπουμε ότι θα αυξηθεί ιδιαίτερα ο χώρος εδώ, σε αυτή τη μικρή δήμο, στην ε, επαρχία του Αλικάντε. Δεν έχει εγκριθεί όμως αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει ο αναφέρον, μια έγκριση έτσι προσωρινή, ας πούμε, από πλευράς Δημοτικής Αρχής, της αυτόνομης όμως αρχής, της, επα... της περιφερειακής αυτής κυβέρνησης είναι αρμοδιότητα σχετικά με το χωροταξικό αυτό σχέδιο. Και ξεκίνησε το 2005 το σχέδιο αυτό, δεν έλαβαν τελικό χαρακτήρα γιατί η αυτόνομη αυτή περιφέρεια δεν ενέκρινε ακόμα αυτό το τελικό χωροταξικό σχέδιο το οποίο δεν ισχύει ακόμα και το σχέδιο το σχετικό ε, γίνεται αντικείμενο ανάλυσης περιβαλλοντικής και με τα πράγματα αναφέρον ακριβώς, αλλά δεν νομίζω ότι όσον αφορά το φυσικό χώρο δεν εφαρμόζεται γιατί δεν επηρεάζεται τα πράγματα για το Natura 2000 και αυτό που είναι σημαντικό είναι η οδηγία πλαισιο για το είδο γιατί όπως λέει ο αναφέρον ακριβώς είχαμε μια έκθεση ε, του Δήμου του Αρμόδιου που έλεγε ότι ήταν δικό αυτό σχετικά με το χορταξ τοξικό αυτό το σχέδιο, γιατί δεν υπάρχουν ε, πηγές ύδατος επαρκής ε, για να εξυπηρετήσουν ακριβώς τις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής αυτής με τον τρόπο αυτό. Και έτσι έχουμε την οδηγία πλαίσιο ας πούμε του ύδατος και όπως είπε ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οδηγία πλαίσιο για το είδωρ πρόκειται για τον ακρογωνίο λίδο πάνω στο οποίο βασίζεται η πολιτική υδάτων ε, της αρχής του 21ου αιώνα από πλευρά πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα και μία αποχρέωση βασική, σημαντική της οδηγίας ε, είναι υδρολογικά ε, πλαίσια κατάλληλα για τις περιοχές αυτές ακριβώς ως ημερομηνία ε, μέσα αυτό το χρονοδιάγραμμα υποχρεώσεων για τα κράτη-μέλη για να εγκριθούν αυτά τα υδρολογικά ε, σχέδια ήταν ε, το, ήταν το 2009 η προθεσμία, εννέα χρόνια μετά από τη θέση σχέση της οδηγίας. Και όσον αφορά την περίπτωση της Ισπανίας δεν εγκρίθηκαν τότε μέσα στην πρόθεσμα τα σχέδια και πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε μια διαδικασία για παράβαση για τα κράτη-μέλη και για την Ισπανία Ισπανία ως αυτά που δεν είχαν εφαρμόσει το σχέδιο αυτό το υδρολογικό. Λοιπόν, σύμφωνα με την οδηγία, αυτά τα υδρολογικά τοπικά ε, σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον έξι μήνες προς έγκριση πριν από την έγκριση αυτή και μετά θα πρέπει να ανακοινωθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία για παρέβαση συνεχίζει απέναντι στην Ισπανία. Ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πρόσφατη 27 Ιανουαρίου συνάντησή της ενέκρινε μια έκθεση αιτιολογημένη κατά της Ισπανίας που ακριβώς είναι η τελευταία φάση πριν να καταλήξει η υπόθεση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς το οποίο νομικά είναι εκείνο που μπορεί να κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που κάποιος δεν σέβεται το κοινοτικό δίκαιο. Στα πλαίσια αυτού του ρολογικού προγράμματο. εκεί προβλέπεται ε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν πηγές υδάτινες για να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες όπως ακριβώς μια παρόμοια χωροταξική οργάνωση και τις νέες ε, κατασκευές ε, που θα γίνουν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν να επαγρυπνούμε για το κοινοτικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αυτή την προσφυγή για παράβαση και έχει προχωρήσει αυτή η προσφυγή κατά της Ισπανίας γιατί δεν σεβάστηκε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο ε, στην περιοχή αυτή όπου υπάρχει και ο Δήμος ε, από το οποίο προέρχονται οι αναφέροντες. Σχετικά με το άλλο σχέδιο του αναφέροντος ε, για το δρόμο τον περιφερειακό στην Δήμο αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι η Οδηγεί επίσης για τις επιπτώσεις και γι' αυτό για ένα δρόμο θα πρέπει να έχουμε μια πρώτα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οποιοδήποτε πελίτης και ο αναφέρον βέβαια μπορεί να αναφέρει τις αντιρρήσεις του, να παρουσιάσει αντιρρήσεις του και να προτείνει άλλε εναλλακτικέ λύσεις σε αυτό το σχέδιο. Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες του αναφέροντας, αυτός ο περιφερειακός δρόμος ούτε αυτός δεν εγκρίθηκε και μέχρι τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα. Και στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μπόρεσε να διαπιστώσει τίποτα προς το παρόν και μια άλλη παράβαση ε, που να μην είναι πέρα από τη μην έγκριση αυτοδρολογικού πλαισίου το οποίο θα πρέπει να επιτρέψει όχι αυτή την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο ο κύριος Ανδρέας Βάρος. Η περίπτωση που αναφέρει ο αναφέρον ακριβώς είναι μια περίπτωση όπου Βρετανοί πολίτες δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ε, σπίτια τους που πίστευαν ότι, θα, ότι είχαν αγοράσει νομίμως την Ισπανία. Η απάντηση που έδωσαν οι Ισπανικές αρχές στην περίπτωση την πρώτη για τα υδρολογικά σχέδια είναι ότι υπήρξε παραβίαση των κανονισμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναλύεται και ως κατάσταση και ίσως θα επιβληθούν κυρώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό βεβαίω δεν αποτελεί λύση για τα άτομα που προσπαθούν να ζήσουν σε αυτά τα σπίτια. Όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο, η απάντηση των αρχών είναι ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο ακόμη δεν έχει εγκριθεί. Και βεβαίως όσοι ζουν σε αυτά τα σπίτια υποφέρουν από τις επιπτώσεις της ε, αρχής του έργου αυτού για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου. Έχουν υπάρξει εδώ και χρόνια παρεμφερείς ε, περιπτώσεις στην Επιτροπή και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα που θα υποχρεώσουν τις Ισπανικές αρχές να προστατεύουν τους πολίτες που ζουν στην Ισπανική επικράτεια στα πλαίσια της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποια και να είναι η ηθαγένειά τους. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί ενδιασμοί για να μιλούμε για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να υιοθετήσουμε την Χαρτή για τα θεμελία δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να συζητήσει οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνει η χώρα τα διάφορα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας υποκριτικός τρόπος να δώσουμε κάποια απάντηση στα άτομα και δεν δίνει πολύ καλή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους πολίτες και τους φορολογούμενους που χρηματοδοτούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανέκλεισε σας, Πρόεδρε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να ενθαρρύνετε την Επιτροπή μας να ζητήσουν από τις Ισπανικές αρχές να απαντήσουν σε όλες αυτές τις αναφορές και μια φορά και για πάντα να επιλύσουν τα προβλήματα που αφορούν την ε, νόμο που πρέπει να ισχύει για τις παράκτιες περιοχές, το νόμο για την ε, ανάπτυξη αστικών περιοχών, ό,τι αφορά την υδροδότηση, οτιδήποτε δημιουργεί πρόβλημα και στους Ισπανούς πολίτες και στους αλλοδαπούς που ζουν στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ομιλητή Χέλμερ. Ευχαριστώ κύριε Εγώ είμαι μέλος του Κοινοβουλίου για 11,5 χρόνια και σε όλη αυτή την χρονική περίοδο έλαβα, λάμβανα επιστολές από άτομα που είχαν ακριβώς τα ίδια προβλήματα όπως αυτά που αναφέρουν ή αναφέροντος. Ε, αγόρασαν ε, σπίτια με σωστά συμβόλαια, καλή πίστη, σύμφωνα με την ε, νομοθεσία και κάποια στιγμή εκδιώκονται με διάφορα τρομερά προσχήματα. Συζητήθηκε πολλές φορές, όπως η κυρία Ανδρεάσεν, πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή μας και δεν βλέπω να υπάρχει πρόοδος. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι κάτι με θυμώνει και με απογοτεύει περισσότερο από το να κάθομαι πάλι και πάλι και να λέω τα ίδια πράγματα στους ε, ψηφοφόρους μου. Λυπάμαι, ξέρω το πρόβλημά σας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα ούτε εγώ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στην απάντηση στην έλλειψη απάντηση που μας παρήχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν ανέφερε καθόλου ή μάλλον σε μία πρόταση μίλησε αρνητικά για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και μίλησε από, για κάποιες σκοτεινές ε, διατάξεις του Natura 2000. Εδώ μιλούμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα να έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία, να έχει μια ιδιοκτησία. Είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι το θέμα της ιδιοκτησίας είναι θέμα ιδιωτικού ε, εθνικού δικαίου. Γιατί πείστε μας λοιπόν κύριε εκπρόσωπο ότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί υπάρχει νομοθεσία για τα ιδιοκτησία ε, των πολιτών και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί μπορεί κάποιο να χάσει την ιδιοκτησία του στι Ισπανικέ Αρχές και δεν μπορεί κανεί να κάνει τίποτε γιατί δεν μπορεί να να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αυτό που λένε αναφέροντος να σταματήσει τι χρηματοδοτήσει προ την Ισπανία η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή αν δεν σταματήσουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ε, διοκτητών οι Ισπανοί. Πιστεύω ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν μια ιδιοκτησία και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως θεμελιώδες δικαίωμα από αυτούς που δεν αναγνωρίζεται, συμπληρωμένες της Ισπανίας και πιστεύω ότι μπορεί για να παγιώσει και να υπερασπίσει αυτά τα δικαιώματα η Κομισιόν κάνει να κάνει. Διότι αυτά τον οποία μας είπε είναι εντελώς απαράδεκτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μακμίλαν Σκότ ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ. 26 χρόνια βρίσκομαι εδώ. 26. Στο πρώτο κοινοβούλιο, στην πρώτη θητεία που ήμουν ευρωβουλευτής, έλαβα μια σειρά επιστολών από ψηφοφόρους μου στο Γιώξια που είχαν αγοράσει ακίνητα στην Ισπανία, κυρίως καμιά φορά και στην Πορτογαλία και έδειχναν μια αυξανόμενη ανησυχία. Τότε είχα οριστεί από την παρούσα Επίτροπη ειδικό εισηγητή για να γράψω έκθεση στην αρχή για διαμεθοριακές ρυθμίσεις ε, στις, ε, στην κυριότητα κινήτων και μετά για το time sharing, το χρονομέρισμα. Ήδη το 1988 μου είχε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπήρχε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυριότητα ακινήτων. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί έχουμε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων με δύο νέα στοιχεία, αφενός τα ε, δικαιώματα για, στην ιδιοκτησία που μας ενδιαφέρει προκειμένου. Υπάρχει και κάποια νομολογία νομίζω της, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που με έχει θέσει υπόψη η νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου και νομίζω ότι τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάψει να αναφέρεται σε παρεμφερή ε, θέματα όπως το περιβάλλον και να έλθει πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Χέλμερ, στα ατομικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα η Επιτροπή μας θα δεχθεί την κυρία Ρέντινγκ, που θα έχει να μας πει κάποια πράγματα για τα νέα δικαιώματα που προβλέπει η συνθήκη. Υπάρχει λοιπόν ένα τρόπος να κινηθεί νομικά προς τα εμπρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχει και ένας πολιτικός δρόμος. Στα 26 χρόνια που έχω συλλέξει εμπειρία στο θέμα αυτό, και κυρίως επρόκειτο βέβαια για Βρετανούς πολίτες που αγόραζαν ακίνητα στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία, σχεδόν αποκλειστικά στην Ισπανία σημειώνονταν προβλήματα. Και δεν είναι αντισπανικό αίσθημα αυτό που εκφράζω εδώ, είναι γεγονότα καμιά φορά είχαν προβλήματα και στην Πορτογαλία. Όχι όμω σχετικά με το νομικό πλαίσιο, αλλά με ορισμένα περιβαλλοντικά θέματα. Είναι πολύ σπάνιο όμω αυτό. Ίσως η κυρία Όκεν έχει κάποια πρόταση ή εσεί, κύριε Πρόεδρε έχετε κάποια πρόταση σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε. Διότι μου φαίνεται ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ένα πλαίσιο δικαίου το οποίο ενδεχόμενα θα αγνοήσει το δικαίωμα υψηλοδιοκτησίας, θα αποτύχει. Και νομίζω ότι η παρούσα επιτροπή πρέπει να είναι και ο μοχλό, ο κινητήρα που θα οδηγήσει προς τα Εμπρό. Κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έξι μήνες μόνο είμαι Ευρωβουλευτής. Και συνεπέρανα ταχύτατα ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται αλλαγή. Το ίδιο διδάσκει εσά η πείρα σα κύριε Σκοτ, που είναι πολύ μακροτέρα βεβαίω. Δεν, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε όμως τέτοια πράγματα να συνεχίζονται. Η οδηγία πλαίσιο για το νερό ίσως είναι ένας τρόπος που μπορεί να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κολυσιεργία της ισπανικής κυβέρνησης στην εφαρμογή των σχεδίων που ασφαλώς αποτελεί φραγμό, εμπόδιο στην τελική διευθέτηση του προβλήματος. Αλλά είναι και το θέμα αυτό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο νόμο για ένα πολίτη της Ευρώπης, άλλο νόμο για άλλους πολίτες της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε συνεκτικότητα και αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι και το κυρίαρχο επιχείρημα εν προκειμένου ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Πρόεδρό μας να εγκύψουν στο θέμα και να βρουν έναν τρόπο σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ε, πολιτών αυτών. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ιτουργκάης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σύντομα σύντομα γιατί οι Βρετανοί φίλοι φίλοι Μακμίλαν και λοιπά, Νομίζω ότι έθεσαν το θέμα όπως ακριβώς έπρεπε όταν είπαν τι μπορούσαμε να κάνουμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ στην Επίτροπη και εξηγούσε αυτά τα διάφορα θέματα που αντιμετωπίσαμε. Είχαμε και αρκετές αναφορές και ισπανικές για χωροταξικά θέματα, για την ακτή, για το περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή και εμείς οι ίδιοι να τα σκεφτούμε εσωτερικά εμείς εδώ. Τι γίνεται με αυτόν τον κόσμο. Πολλές φορές ε, ε απασχολούν ακριβώς, ε, δεν θα πρέπει να τους ξεγελούν και τους ξεγελάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από αυτά που μπορούν να γίνουν κανονικά εδώ. Γιατί έχουμε όρια εδώ που είναι της δικής μας Επίτροπης. Αυτοί είναι κανόνες του παιχνίδιου και προσπαθούμε βέβαια. Γιατί το λέω αυτό. Όταν ε, αντιθήκαμε οι συντονιστές και ε, ζητήσαμε και στην Ισπανική κυβέρνηση είχαμε μια κρόση για θέματα χωροταξικά, των ακτών, διάφορες ε, αναφορές που αφορούσαν κυρίως τις ισπανικές περιπτώσεις, αλλά εμείς από την Επιτροπή Αναφορών βλέπουμε ότι έχουμε ξεκινήσει ένα δρόμο μια πορεία με επιστολές όπως είπαν οι συνάδελφοι και από τους συντονιστές ας πούμε στον ε, Ισπανό διαμεσολαβητή και να μας μπορέσει να μας εξηγήσει και να μας πει ποια είναι εντύπωσή του για αυτές τις περιπτώσεις και επίσης δρόμους και πορείες στα πλαίσια ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλες επιτροπές όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος ή την Νομική Επιτροπή να μπορεί κανείς ε, να βασιστεί κάπου περισσότερο για αυτές τις αναφορές ε, να έχουν περισσότερο βάρος εκεί. Μερικές φορές με εκπλήσει κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε αυτές τις ισπανικές περιπτώσεις ε, κάθε τόσο εδώ και έχουμε 10, 15, 20 ισπανικές αναφορές και συνεχώς μιλάμε για την Ισπανία, πώς έχει αρνητικά η κατάσταση, εντάξει θα μπορούσε να βελτιωθεί, πάντα το είπαμε, η Ισπανικός νόμος και σχετικά με όλα αυτά και από πλευράς του κόμματός μου πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί αυτό σχετικά με τις ακτές κλπ. Και αν κερδίσει το ΕΛΚ ε, μεθαύριο θα καταβάλουμε προσπάθεια βέβαια να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί για τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά κύριε Πρόεδρε αυτό που ισχύει είναι ότι γύρω-γύρω περιφερόμαστε. Πολλές φορές ακούμε, ακούμε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι οι Βρετανοί κυρία, και, και, και λοιπά. Και εγώ μπορώ να το πω και άλλοι συνάδελφοι μπορώ να το πούν ότι μπορούμε να δούμε ακριβώς το, τις ενέργειες και να είναι φωτοαντίγραφα. Τα ίδια λέμε, τα ίδια παραλαμβάνουμε, τις ίδιες θέσεις ακολουθούμε. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Αυτή είναι η θέση μας. Εντάξει, αυτό είμαστε σαν Επιτροπή Αναφορών στιγμή λοιπόν που δεν είμαστε σε θέση να ακούσουμε, να, να ακουστεί αυτό που λέμε εμείς, δυστυχώς, δυστυχώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτήν την Επιτροπή. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία να έχει το λόγο και μετά καλό σύντομα όμως γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε έτσι με την μυρίσια διάταξη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι σύντομη. Ε, ε, συμφωνώ με τον κύριο Ιτουργκάης συχνά ότι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο Βρετανοί πολίτες. Στην έκθεσή μου είχαμε πολίτες από όλη την Ευρώπη. Και οι περισσότεροι μάλιστα ήταν Ισπανοί. Το θυμίζω αυτό. Έχουμε την άμεση δυνατότητα, όπως είπα στην έκθεσή μου, να δούμε και τα οικονομικά. Αλλά τι έγινε όταν συζητήσαμε τελευταία φορά, την, όταν συζητήσαμε με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Προσπάθησε να αποφύγει η Επιτροπή Προϋπολογισμών την σχετική ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Μπήκε στην άκρη διότι είχε υπάρξει συμβιβασμός. και θα τα μείωνε τα χρήματα, θα μείωνε τα κονδύλια. Είμαι βέβαια ότι κάποιος το έκανε. Εν πάση περιπτώσει είχα την αίσθηση αυτή. Ε, ίσως έχουμε περισσότερες δυνατότητες μέσω του οικονομικού. Δεν είναι μόνο το θέμα του χάρτη. Θα σας έλεγα όχι. Μην βάλετε θέμα χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω στο άρθρο 11 της συνθήκης λέει καθαρά ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν επεκτείνει την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στις χώρες μέλη. Το λέει καθαρά. Και το επιχείρημα το χρησιμοποιεί αυτό διαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορεί, δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα ο χάρτης. Αλλά έχουμε το άρθρο 7. Να είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε, όταν επικαλούμαστε το άρθρο 7. Γιατί πρέπει να είναι δραματική κατάσταση για να επικαλεστεί κανείς το άρθρο 7. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ να χρησιμοποιηθεί για θέματα ελευθερία τύπου στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, τέτοια πράγματα. Αλλά όχι να, μην είναι η κατάχρησή του όμω, είναι σημαντικό αυτό. Το άρθρο 7 τώρα μα δίνει τη δυνατότητα στην προηγούμενη συνθήκη το μόνο που, σας, το μόνο που έμενε ήταν εκτελέσει στην αυγή. Και αν δεν έχει κανεί τι εκτελέσει στην αυγή δεν έχει τίποτα. Όλοι μπορούν να πούν, και ο Κομισιόν μπορεί να πει ότι κάτι πάει στραβά εδώ, κάτι πάει σοβαρά στραβά. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Είναι σαν να τους δείχνετε μια κίτρινη κάρτα. Μετά να δούμε αν αυτή η κίτρινη κάρτα πραγματικά αποδίδει. Και νομίζω στα τέσσερα πέμπτα των χωρών μελών, πολλά τέλο πάντων, μπορεί να σηκώσει, να δείξει την κόκκινη κάρτα. Που σημαίνει ότι θα προβεί σε σοβαρές έρευνες η Επιτροπή διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και μετά ακολουθεί αν δεν γίνει τίποτα εκτέλεση την αυγή. Πάντως έχουμε πλησιάσει να κάνουμε κάτι εάν ε, επικαλεστούμε το άρθρο 7. Όπως κάναμε και με την εκθεσή μου που ήταν νομίζω το άρθρο 6 της προηγούμενης συνθήκης νομίζω να το εξετάσουμε σοβαρά, τέλος πάντων. Και το τελευταίο μου θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με την ε, νομοθεσία περί ακτών, που εκεί τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Ο νόμος εντάξει είναι, αλλά δεν εφαρμόζεται καλά. Αν εφαρμοζόταν ο νόμος, η Ισπανία σήμερα θα ήταν μια κούκλα, αλλά έχει εφαρμοστεί με πολύ αυθαίρετο τρόπο ο νόμος αυτός. Μην αναμίξετε το θέμα αυτό τώρα εδώ με το νόμο περί ακτών. Το τονίζω αυτό. Είναι ένα θέμα που η Κομισιόν ακόμα δεν το έχει ανακαλύψει. Ότι έχουμε το άρθρο 7 δηλαδή στη διάθεσή μας. Κύριε Πιτουργκάιτ, ναι, η Επιτροπή Αναφορών είναι αυτή στην οποία απευθύνονται οι πολίτες έρχονται εδώ με δάκρυα στα μάτια και ασφαλώς και πρέπει να τους σεβαστούμε. Και από όλα τα μέρη έρχονται. δεν είναι κυρίως δική μου ψηφοφόρη, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους. Ευχαριστώ κύριε Άουκεν. Παρακαλώ να είστε σύντομοι συνάδελφοι, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Κύριο κύριος Μαρτίνε. Θα είμαι σύντομος. Ε, υπάρχουν πράγματα που είπαν άλλοι συνάδελφοι, όπως είπε η κυρία Άκεν, σχετικά με το σεβασμό αυτού του χάρτη. Είναι απόλυτα σωστό η χρησιμοποίηση και λοιπά Η χρήση. Αλλά μιλήσαμε αρκετές φορές για την συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι που κόσμος συνάδελφοι που είναι ριζικά αντίθετοι για να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη σύμβαση από το Σύμβουλο της Ευρώπης που προερχόταν. Ε, χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν συνάδελφοι που ε, αναφέρονται ακριβώς σε αυτή τη σύμβαση, έτσι. Αυτή η σύμβαση, από ό,τι γνωρίζω, κάτι το, παραμένει κάτι το ανοιχτό για να μπορέσει κανείς και να καταγγείλει το γεγονός στον αρμόδιο οργανισμό, στον αρμόδιο φορέα, οποιοδήποτε πολίτης που προέρχεται από μια χώρα, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, με συγχωρείς, με συγχωρείς Εντουάρντα, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να καταγγείλει κάτι μπροστά στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το οποίο θα αποφασίσει. Αυτό το δικαστήριο πέρα, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. οποιοδήποτε επαναλαμβάνω, πολίτης ε, από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, μπορεί από τη στιγμή που θεωρήσει κάτι ότι είναι παραβίαση αυτού της, αυτής της μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο, γι' αυτό υπάρχει αυτό το δικαστήριο και και να δούμε ακριβώς ε, τι γίνεται και ότι υπάρχει δυνατότητα δικαστικών αποφάσεων που είναι δεσμευτικές χωρίς να έχουν ε, δυνατότητα έφεσης. Εδώ μιλήσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώς και βέβαια ορισμένο σε αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα ιδιωτική ιδιοκτησία είναι εκείνο που, που να πιστεύει ότι υπερισχύει οποιοδήποτε άλλο. Ορισμένοι δεν το πιστεύουμε αυτό, έτσι. Ορισμένοι θεωρούμε ότι η, ιδιωτική, ιδιοκτησία έχει τη σημασία τη βέβαια, αλλά δεν είναι ανθρώπινο δικαιώματα που υπερισχύει απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα και ότι υπάρχουν δικαιώματα και μάλιστα συλλογικά, ομαδικά, που υπερισχύουν νομίζω με απέναντι στο δικαίωμα ατομική διοκτησία διαδικασίες, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση. Ε, σύμφωνοι παλιότερα σε άλλους ε, όπως ο Ήρβιν, η Ομεριμέ, στην ε, διηγήματα της Αλάμπρας έλεγαν ας πούμε ότι τι γινόταν, ε, τα υποστήριζαν αυτά σε παλιότερα διηγήματα παλιότερων αιώνων, αλλά αυτά είναι ξεπερασμένα τώρα πια. Εγώ βλέπω αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κ. Σοτοργάη ότι η αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής Αναφορών πια είναι βέβαια σε κάποιες στιγμές ε, ίσως ε, καταλήξει σε τείχος των δακρύων, σε τείχο των δακρύων. Και Ορισμένοι ραπονιούνται, έρχονται εδώ, τους ακούμε και βλέπουμε ότι βλέπουμε πολλές και πάρα πολλές αναφορές, παραμένουν ανοιχτές και τότε καταπιέζονται όλα αυτοί, αισθάνονται άσχημα. Και μάλιστα και αρκετοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν αυτή η καταπίεση είναι στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα του καθένα να αισθάνεται καταπιεσμένος. Ε, εντάξει, τέλος πάντων, ε, μερικές φορές και εγώ αισθάνομαι καταπιεσμένος έτσι το λέω αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Η Ισπανία είναι μια χώρα δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα που υπάρχει ε, υποδειγματικό σεβασμό των ανθρωπίνων Όχι, τέλο πάντων, εδώ και για 40 χρόνια δεν γινόταν αυτό. Όχι όμω τη ιδιωτική ιδιοκτησία. Η Ισπανική δικτατορία, όπω και η Χιλιανή, όπω οι διάφορε δικτατορίε που είδα εδώ και εκεί στο δυτικό κόσμο, αυτέ όλε διατηρούσαν το δικαίωμα τη ιδιωτική ε, ατομική ιδιοκτησία, ήταν από τι βάσει ε, ε, των ε, καθεστώτων τους. Θεωρώ λοιπόν εντάξει ότι ε, σεβόμαστε στην Ισπανία τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά ήθελα να το πω όχι μόνο στους συναδέλφους που πήραν το λόγο πάνω σε αυτό μεμονωμένα αλλά γενικότερα θα πρέπει οι ίδιοι να αναρωτηθούν γιατί τώρα πέρα από αυτές τις συμβάσεις, από αυτές τις επιστολές ε, τις συζητήσεις ε, είχαμε Βρετανούς Βρετανούς και Γερμανούς και Αυστριακούς πέρυσι που αγόρασαν σπίτια στην, ε, στην, Ισπανία περισσότερες από ότι, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι άλλα χρόνια. Πολίτες ακριβώς σε αυτόν τον χώρο που μόλις ανέφερε, δεν ξέρω, μήπως δεν είναι καθόλου μα καθόλου κατά Τοπισμένοι είναι μαζοχιστές, θέλουν να υποφέρουν και πάνε και αγοράζουν σε μια χώρα που όπως λένε εδώ πέρα είναι ότι παντού τους κατακλέβουν ε, στις ιδιοκτησίες τους. Εγώ έχω στο Αλικάντε μια μια, ένα σπίτι και είμαι σε ένα χώρο που είμαι μοναδικός Ισπανός. Παντού είναι Ισπανοί, ε, παντού είναι Γερμανοί, Γάλλοι, ένας Ελβετός εδώ και εκεί. Είμαι μόνο εγώ Ισπανός είπαμε, έτσι. Και κανείς δεν είναι που να παραπονιέται ότι τον κατάκλεψα τον Αταλό. Είχε καμία περίπτωση από αυτές. Άρα λοιπόν δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και ατασταλίες και διάφορα παρατράγουδα. Υπάρχουν και βέβαια παρόμοιε περιπτώσει θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε. Μην δίνουμε όμω την εντύπωση ότι το σύνολό τη η Ισπανία είναι μια χώρα που καταπι... παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, αυτό είναι έτσι κάτι το παραμορφωμένο, γκροτέσκο είναι και παρόμοια όλα αυτά που επαναλαμβάνονται εδώ όχι, ε, δεν είναι υπερβολή να αυτό το λέμε αυτό, γιατί και στη Λονδίνο, ας πούμε, είναι για 90 χρόνια κάνεις ε, κάποιος ε, κύριος, δεν είναι υπερβολή ότι αυτό που λέμε ότι γίνεται το ένα Βασίλειο και ότι είναι εις βάρος του κόσμου ακριβώς μόνο και μόνο επειδή κάποιος είναι κύριος ενός ε, ε κύματος για 90 και μόνο χρόνια. Θα πρέπει να προσέχουμε κάθε περίπτωση εδώ. Τέλος πάντων θα πρέπει κάπως να σεβόμαστε το κάθε κράτος μέλος ακριβώς τα πλαίσια αυτού του σχεδίου γιατί η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που μας ενώνει βέβαια και να δούμε τώρα με τους μηχανισμούς αν ε, σημειώνεται ή όχι παραβίαση αυτών ε, και με τις κοινοτικής νομοθεσίας. Νομίζουμε ότι όλα αυτά ισχύουν, υπάρχουν και μας βοηθούν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι δια εκθέσεις ε, θα διατηρηθούν ανοιχτές για να εργαστούμε πάνω σε αυτές, να δούμε ανάλογα βέβαια και με τις αρμοδιότητες επιτροπής μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ να σας πω κάτι, ότι έχουμε πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα χρόνου τώρα εδώ. Έχουν ζητήσει το λόγο η κυρία Βέτμαν, Γκουτιέρε, Ουστινά, Μπουστινάρο, Ανδρέας και Μακμίλαν όλοι αυτοί και έχουμε στη διάθεσή μας μόνο 12 λεπτά. Θα πρέπει μετά να, θα πρέπει να σεβαστούμε την ημερήσια διάταξη γιατί δεν θα μπορέσει να έρθει εδώ ο εκπρόσωπος της Επιτροπής το απόγευμα. Παρακαλώ ένα λεπτό το πολύ ο καθένας έτσι, άντε 50 δευτερόλεπτα <laughs> όπως και στην Ολομέλεια το ίδιο θα πρέπει να σεβαστούμε. Και εντάξει παρακαλώ μην επαναλάβουμε πράγματα Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση, επαναλαμβάνομαι. Θα ήθελα να υποβάλω μια πρόταση εγώ. Η ε, κυρία Βέτμαν. Αυτό θέλω να βάλω σαν πρόταση εγώ. Βέτμαν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν θέλω να μιλήσω για δικαιώματα κυριότητας ή ατομικά δικαιώματα ή ε, χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων που νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Θα έλθω σε ένα θέμα, την αρμοδιότητα της Επιτροπής, της Κομισιόν δηλαδή. Διότι τον Οκτώβριο 2003 εξέδωσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή τότε θα ετίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Νίκαιας, και για το άρθρο 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, λέει εκεί λοιπόν η συνθήκη της Νίκαιας δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου, να αναλαμβάνει δράση και επομένως νέα αρμοδιότητα για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα η αρμοδιότητα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ήδη από το 2003 και τώρα που έχει πλέον τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και επομένως έχει γίνει και ο χάρτης θεμελιών δικαιωμάτων <clears throat> εξαναγκαστό δίκαιο, γιατί δεν υπάρχει πλέον αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα θέμα που οποίο πρέπει να τεθεί. Ευχαριστώ κύριε Βέτμαν. Κύριε Γκουτιέρες. Ένα Η Ευρώπη όπως έπρεπε και το λέμε με απόλυτη σαφήνεια, ποτέ δεν έκανε τίποτε υπέρ των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Βλέπουμε όμως ότι η είχαμε στην περίπτωση των ε, κρατών της Ανατολικής ε, ε, Ευρώπης ότι υπήρχαν τρομερά προβλήματα διαφθοράς, διαφθοράς και θέματα ε, αγοραπολισιών και επιστροφής διοκτήσεων. Αναφέρομαι στην κροτή. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι στην ε, βόρεια η Ισπανία όπου υπήρχαν, ε, όπου θέλαμε να μην γίνει τίποτε και υπήρξε μετά από κάποια χρόνια εκ μέρους του Δημάρχου κάποια απόφαση να γκρεμιστούν αυτό και άλλα ωραία σπίτια για να χτιστούν άλλα. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι αντίθετη προς την οποιοδήποτε νομοθεσία την ισπανική που δεν ορίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα των ιδιοκτητών. Θεωρώ ότι θα πρέπει Όπω είπε και ο κύριο Μακμίλα να δούμε με σαφήνεια τα πράγματα και να τα διαχωρίσουμε. Όταν υπάρχει πρόβλημα παραβίωσης της κοινωτικής νομοθεσίας να ασχοληθούμε. Στην Ισπανία υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και πολλές φορές γίνονται καταχρήσεις. Και πρέπει να πω ότι όντω έχει αποδειχθεί ότι για θέματα ε, ενδιαφέροντος του κράτους πραγματικά πλήττονται πάρα πολλά δικαιώματα ιδιοκτητών. Πολλές φορές όμως ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει και εκ μέρους κάποιων ιδιοκτητών σωστά, διότι για να εξοικονομήσουν κάποια έξοδα δεν περνούσαν από την νόμιμη οδό, πήγαιναν μόνο σε ένα συμβολιογράφο και παίρνουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. όπως είπε ο κ. Μακλίν, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σωστά ποια είναι τα πράγματα και να κάνουμε διαχωρισμό. Σύντομα, ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ, πρώην. Θα μιλήσω ρουμάνικα. Πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποια είναι τα προβλήματα για να δούμε ποιες είναι οι λύσεις που θα δώσουμε. Θα δούμε, πρέπει να δούμε επίσης ποια είναι τα προβλήματα που ανέφερε η Επιτροπή και να λάβω υπόψη και το ότι δεν υπάρχει αντίδραση μέσα των Ισπανικών αρχών. Πολύ συχνά και για τις αναφορές 8 έως 12 γίνεται λόγος για σχέδια τα οποία θα εφαρμοστούν, που ακόμη δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τα σχέδια αυτά έχουν εγκριθεί. Προτείνω λοιπόν η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Η Επιτροπή επίσης θα πρέπει να κοινοποιήσει στις ισπανικές αρχές την όλη κατάσταση και να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για τους φακέλους αυτούς και να ζητήσει η Επιτροπή μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρακολουθεί εκ του καλύτερα τις εξελίξεις είναι σαφές ότι είναι απαράδεκτο να λέγεται ότι είναι διεφθαρμένο κράτος η Ισπανία. Και δεν θα πρέπει να λέμε όπως κάποιοι συνάδελφοι ότι είναι ληστρικό κράτος η Ισπανία. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους ε, παρατηρήσεις για ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα, όποια και να είναι η κυβέρνηση. Και ας μην κάνουμε πολιτικές θεωρήσεις και ας μην αναφέρουν κάποιοι συνάδελφοι τι έκαναν οι προηγούμενες ε, ισπανικές κυβερνήσεις της δεξιάς. κυρία Αντρίσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς θέλω να πω σε σχέση με όλες αυτές τις αναφορές και τις παρεμφερείς που έχουν φτάσει στην Επιτροπή μας τις τρεις-τέσσερις τελευταίες ε, δεκαετίες, το κλειδί είναι, είναι ε, νόμιμο και σωστό να συνεχίζει να χρηματοδοτεί οι ευρωπαϊκές περιοχές που κάνουν τέτοιου είδους ε, παραβιάσεις. Κύριε Τουργάης, ίσως τα θέματα αυτά θα πρέπει να πάνε στην Επιτροπή Προπολογισμών και ελέγχου των προπολογισμών. Να είστε σίγουροι ότι αν φτάσουν, εγώ θα μπλοκάρω τη χρηματοδότηση μέχρι να ευρεθεί λύση. Τώρα, στον κύριο Μαρτίνε, όσον αφορά τι αρμοδιότητε του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να πω ότι το δικαστήριο δεν ε, παίρνει δεσμευτικέ αποφάσει, απλώ κάνει κάποιε συστάσει. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Μακμίλαν. για αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο. Να απαντήσω τον κύριο Μαρτίνες. Τα συμβατικά ανθρώπινα δικαιώματα του 1949, πρωτοκόλλο 1, περιλαμβάνεται εκεί το δικαίωμα ε, ιδιωτικής κυριότητας, αλλά δεν το έχει υπογράψει η Ισπανία αυτό το πρωτόκολλο. Και άλλες χώρες βέβαια. Και επομένως δεν εφαρμόζεται στην Ισπανία. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντα θέλω να διατηρηθεί ανοιχτή η ε, αναφορά αυτή και να εξετάσουμε εμεί ως Επιτροπή Αναφορών εάν θα ζητήσουμε επίκληση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων να δούμε στην, στον τομέα αυτό ποιες αρμοδιότητες έχει εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, επιβολή των διατάξεων του χάρτη. Η Κομισιόν. Μια στιγμή, μια στιγμή. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Φύγαμε από τα θέματα του νερού, που ήταν δραματικά βέβαια, και ήρθαμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυρία Άουκεν και ο κύριος Μαρτίνες μας θύμισαν σωστά τους περιορισμούς εφαρμογής του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβάνονται στο άρθρο 51, αλλά επειδή μου ζητήσατε να είμαι σύντομος, θα επανέλθω σε δύο μόνο σχόλια που έγιναν σχετικά με τον προϋπολογισμό. Υπενθυμίζω στην κυρία Άουκεν τι έγινε ακριβώς στην προηγούμενη, στο τέλος της προηγούμενης θητείας. Είχε προταθεί η διακοπή της καταβολής κονδυλίων των διαρθωτικών ταμείων στην Ισπανία, μέχρι ότου υπάρχει διαβεβαίωση από τι αρμόδιε αρχέ ότι έχουν σταματήσει οι πρακτικές αυτές. Πέρασε από... Έφτασε μέχρι την Ολομέλεια, αλλά καταψηφίστηκε η πρόταση αυτή στην πρώτη ανάγνωση. Το θυμούμε καλά γιατί ήμουν παρόν και μου είχε φανεί πάρα πολύ σημαντικό γεγονό αυτό. Δεύτερο, για την κυρία Βέτμαν αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην πραγματικότητα η ανακοίνωση εκείνη, που δεν αποτελεί νομικό κείμενο, αυτό που είχε ως αντικείμενο ήταν να προσφέρει ορισμένα επιχειρήματα για την ίδρυση του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υπάρχει τώρα. Σε πολλές από τις συζητήσεις αυτές, ίσως θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια για τις διαβουλεύσεις τη η Επιτροπή Αναφορών, ακριβώς από τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Ο αναφέρον έχει το λόγο. Τελευταίος. Πριν από την πρόταση. Πώς να απαντήσω σε όλα όσα άκουσα σήμερα. Θα πω μονάχα ότι ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πελάτης της Ευρωβουλής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Είμαι απογοητευμένος από το γεγονός ότι το όργανο σας θεωρεί ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να απαιτήσει από μια χώρα μέλος που λαμβάνει τόσες επιδοτήσεις να συμμορφώνεται με θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ Σίγουρα παραμένει ανοιχτή αναφορά για όλους αυτούς ε, τους λόγους και για τις πληροφορίες επίσης για την τολιμή έκθεση και για την διαδικασία παρεμβάση όπως και αυτό ακριβώς που, ήταν, που έγινε πέντε μέρες πριν ε, για το είδωρο. Εγώ θα ήθελα να αποβάλει μια πρόταση σαν επιτροπή να απευθυνθούμε στην Ισπανία για να, να ζητηθεί από την Βαλένθια την περιφερειακή κυβέρνηση να μας ενημερώσει για το σχέδιο τους, αυτού του Δήμου, το οποίο εγκρίνεται, εγκρίθηκε το 2009 από το Δήμο ακριβώς, αλλά η χωροταξική αρμοδιότητα είναι της αυτόνομη κυβέρνησης, δηλαδή της Βαλένθια και σίγουρα συμφωνώντας με την ανησυχία που εκφράστηκε και από τον αναφέροντα και από δική σας πλευράς να απευθυνθούμε ακριβώς στην περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια και να μπορέσουν έτσι να μας εξηγήσουν εκείνοι πώς έχει κατάσταση με αυτό το γενικό σχέδιο που εγκρίθηκε το 2009 αλλά που προς το παρόν δεν έχει προωθηθεί. Και από τη στιγμή που θα έχουμε τη σχετική πληροφορία θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα. Παρακαλώ στις 4.30 να σας υπενθυμίσω ότι η Επίτροπος Βίβια Ρέντινγκ Αντιπρόεδρος Επιτροπής θα είναι παρούσα για να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα των πολιτών. Ευκαιρία δεν είναι μαζί της να μπορέσουμε να δούμε αυτές τις γενικές περιπτώσεις. Σίγουρα θα πρέπει να σας πω ότι εδώ όταν αντιμετωπίζουμε παρόμοια θέματα που έχουν να κάνουν με κράτη-μέλη δεν σημαίνει ότι αμφισβητούμε αυτή την νομιμότητα. Είναι ειδικέ περιπτώσεις, συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές οι υποθέσεις που αφορούν ε, τα κράτη-μέλη. Ασχοληθήκαμε με τη Βουλγαρία, ασχοληθήκαμε με την Ισπανία. Σίγουρα, δυστυχώς ε, είναι εκτεταμένη χώρα η Ισπανία, είναι μια χώρα βέβαια ευχάριστη για να ζει κανείς εκεί. Γι' αυτό πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, τα βουνά της πόλης σακτές επιλέγουν για να ζήσουν εκεί και είναι ένα φιλόξενο κράτος. Ισπανία μπορεί κανείς να ζει ευχάριστα εκεί, άρα λοιπόν παρουσιάζονται τελικά προβλήματα εκεί. Έτσι. Στα πλαίσια αυτής της συμβίωσης όμως εδώ ε, περνάμε το σημείο αυτό λοιπόν, τελειώνουμε και αν έχουμε χρόνο για να δούμε... Για να δούμε. Έχουμε πολύ ο χρόνο, μήπως θα μπορούσαμε να περάσουμε να έρθουμε στο σημείο 8 που το είχαμε παρακάμψει το σημείο 8. Είναι η 437 του Χωσή Αντώνιο Μοδοκράου Εξονόμαστε τη την Κομισιών Προρίο σχετικά με τη ρήπανση του ποταμού Σεγούρα στην περιφέρεια Μόρθια. Δεν είναι εδώ αναφέρον. Ο εκπρόσωπος τη Επιτροπής Ευρωπαϊκής όμως έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτές τις δύο εκθέσεις, ε, δύο αναφορές, έχουμε δύο είδη προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα για τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία των υδάτων ε, κατά μόλις και λοιπά από νητρικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και επίσης ε, το θέμα του σεβασμού της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ε, νερά των πόλεων και ακόμα για τη ρήπαση του ποταμού Σεγούρα στην περιφέρεια Μούρθια. Εμείς ολοκληρώσαμε και ολοκληρώνουμε σε ορισμένε περιπτώσεις με τα αντικείμενα αυτών των αναφορών ε, έρευνες για να δούμε για τον σεβασμό ας πούμε της οδηγίας για ε, αζωτούχα λοιπάσματα και η Επιτροπή ξεκίνησε μια σχετικά με τη διαδικασία για παράβαση, για παραβάσεις ε, σχετικά με τα ύδατα και αυτό έχει να κάνει όμως με την Μούρθια. Γιατί, γιατί βάσει της σχετικής ε, διαδικασίας από την Επιτροπή ε, οι αρχές ε, τον Ιούνιο του 2009 είδαν ποιες ε, πρόσεξαν να δουν ποιες είναι οι τελευταίες περιοχές που είναι ευαίσθητες στην χρήση ε, αζωτούχων λιπασμάτων για να επιλύσουν το πρόβλημα και σε σχέση με ε, την υπόλοιπη αιτιολόγηση αυτής της διαδικασίας για παράβαση ζητείται η υιοθέτηση προγράμματων δράσεων για αυτές τις περιοχές και ακριβώς ε, στην περιοχή της Μούρθια προχώρησαν εκεί σε προγράμματα προστασίας που ικανοποιούσαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 δηλαδή σχετικά με την οδηγία για τα ζωτού χάλατα δεν υπάρχουν περιπτώσεις κρεμής σχετικά με την περιοχή της Μούρθια ενώ για το δεύτερο σημείο για την έκθεση αυτή για τις υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όπως ενημερώσαμε εδώ την Επιτροπή αρκετές φορές, η Επιτροπή ξεκίνησε διάφορες διαδικασίες για παράβαση κατά της Ισπανίας με όλες τις αυτόνομες περιοχές που έχουν σχέση με αυτό. Αλλά μέχρι τώρα για τον σεβασμό αυτών για τα απόλυτα και στις περιοχές αυτές που είναι στο ποταμό Σεγκούρα στην περιφέρεια Μόρθια μπορούμε να πούμε ότι λήφθηκαν τα μέτρα και σέβονται την οδηγία αυτή. Γιατί το διευκρινίζω. Δεν είναι πέρα από αυτήν την ε, σεβασμό ε, δεν έχει να κάνει με το σεβασμό άλλων περιοχών, αλλά εδώ ε, είναι για περιοχές που ρίχνουν τα νερά τους στον ποταμό Σεγκούρο. Υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν το πρόβλημα και των ε, αζωτούχων λιπασμάτων και από τη γεωργία και την επεξεργασία αποβλήτων υδάτων. Ε, νομίζουμε ότι βάσει των πληροφοριών έχουν λυθεί το προβλήματα σχετικά με τον ποταμό αυτό στην ε, Μούσια. Παρακαλώ. Ναι, το είπε ήδη η Επιτροπή ότι είναι το 2001 η καταγγελία αυτή. Το 2010 έχουν λυθεί τα προβλήματα από τα περιφερειακά ταμεία ε, λύσαμε το πρόβλημα και βλέπουμε αυτόν τον καρπό των προσπαθειών βέβαια και μετά από τη ρύθμιση αυτή μπορέσαμε να βοηθήσουμε αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι δεκτή αυτή η αναφορά αλλά τελικά τι γίνεται, εδώ μας κάνουν να χάνουμε χρόνο και σε εμά και σε όλους. Ε, εδώ έχουμε μια καταγγελία, εντάξει, θα μπορούσαμε να την είχαμε υποστηρίξει τότε. σχετικά με, το, με τα σχέδιά τους ε, έχουν να κάνουν με την οδηγία αλλά δεν προχώρησε γιατί οι περιφερειακές ε, κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι είναι περιφερειακή αντιμετώπιση αυτή. Είναι ε, δύσκολο το θέμα. Υπάρχουν καταγγελίες, θα πρέπει να υποστηρίξουν την κεντρική κυβέρνηση για να αντέξει την πίεση από τις αυτόνομες περιφέρειες, τίποτα άλλο. Διάφορες όμως καταγγελίες έτσι ξεπερασμένες ε, δεν θα πρέπει να γίνουν δεκτές γιατί μας κάνουν και χάνουμε το χρόνο μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, από τις δύο παρεμβώσεις και τις Επιτροπές Επιτροπής και της κυρίας Γκουτιέρης έχει ε, κλείσει το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν περνάμε στο σημείο 12, το επόμενο σημείο που έχει να κάνει με την αναφορά 584 του Πέντρο Κουέβας Κουέτο, Ισπανικής Σταγένεια, σχετικά με την επέκταση του αυτοκινοδρόμου Α8 στην περιοχή της Καντάβριας. Επιτροπή, ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, η αναφορά αυτή έχει να κάνει με τη διέλευση από την περιοχή Καντάμπρια από στο βορρά της Ισπανίας, η Α8, Α8 και πάει από το Λιάνες ε, στην Αστούριας μέχρι τον Κέρα στην ε, Καντάμπρια σε άλλη περιοχή δηλαδή. Και εδώ ε, επηρεάζεται το περιβάλλον και κυρίως το ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Ε, τα σπήλαια του καταμετέρω στο Λιάνες ε, που σύμφωνα με τον αναφέροντα θα επηρεαστούν αυτά τα πράγματα αρνητικότατα από το πέρασμα αυτού του αυτοκινητόδρομου. Οι υπηρεσίε Επιτροπή εξέτασαν τα διάφορα επιχειρήματα του αναφέροντος και ε, όσα είπε εκείνο και όλα τα προηγούμενα που είχαν σημειωθεί για το θέμα αυτό, για την περίπτωση αυτή. Όσον αφορά το δίκαιο για το περιβάλλον, η οδηγία η σπουδαιότερη είναι των επιπτώσεων, 85 η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε διάφορα δημόσια προγράμματα και ιδιωτικά, σύμφωνα και με το παράδειγμα 1 και 2 της οδηγίας. Επίσης, και τα σχέδια για αυτοκινοδρόμους αναφέρονται στο παράδειγμα 1 της οδηγίας και η πραγματοποίηση ακριβώς μιας διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων είναι κάτι το ε, απαραίτητο δεσμευτικό. Σχετικά με το άρθρο 3 της οδηγίας επίσης για το περιβάλλον έχουμε πολλούς παράγοντες εκεί όπως και η πολιτιστική κληρονομιά που συμπεριλαμβάνεται. Άρα λοιπόν μιλάμε και τις επιπτώσεις πάνω στη φύση αλλά ταυτόχρονα αναφερόμαστε και στην πολιτιστική ή ιστορική κληρονομιά. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη ήταν γνώστοι στο θέμα αυτό γιατί ήδη υπήρξε παράπονα το 2005 τότε είχε κλείσει η υπόθεση από την Επιτροπή γιατί δεν πιστοποίησαν μία, δεν διαπίστωσαν μία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Το 2009 ακούσαμε νέα παράπονα σχετικά με το ίδιο αυτό πρόγραμμα και πάλι δόθηκε τέλος έκλεισε η υπόθεση αυτή από την ώρα σε αυτό το σχέδιο είναι μια σαυτοκινοδρόμος 22 περίπου χιλιόμετρων και είχαμε μια διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον και έγινε μια δήλωση που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 25 Ιανουαρίου του 2006 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής που στάθηκε στην Επιτροπή σας εδώ. Εδώ αυτό το σχέδιο με αρκετέ διαφορές και αντιδράσεις είχαμε δύο περιπτώσεις εκτίμησης επιπτώσεων, το μία το 1993 και μία άλλη δεύτερη το 1996. Γιατί αυτές οι δύο διαφορετικές διαδικασίες για τις επιπτώσεις περιβάλλον. Ε, χάρη σε αυτές όμως άλλαξε το σχέδιο και προσπάθησαν να βρουν εναλλακτικέ λύσεις που θα σεβόταν περισσότερο το περιβάλλον σε από άλλες περιοχές σύμφωνα και με το σχέδιο Natura 2000 και να υπάρξουν όσο γίνεται ελευθερότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον ότι από πλευρά πολιτιστικών οργάνων ε, και περιβάλλοντος επίσης έγινε διαβούλωση με αυτές τις αρχές για να πούν την απόψή τους. Και ακόμα κάτι πρόκειται για ένα σχέδιο που υπήρχαν διαφορές αντίδρασεις έντονες και υπήρξαν και προσφυγές στα ισπανικά δικαστήρια και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ταυτόχρονα υπάρχει μια διοικητική προσφυγή εκκρεμή μπροστά στο εθνικό όργανο και δεν μπορούσαν να, διαπιστ... δεν να διαπιστώσουν μια παραβίωση τουλάχιστον υπηρεσία της Επιτροπής και έτσι υπήρξε μια εκτίμηση σίγουρα επιπτώσεων αλλά αυτή η ανάλυση ήταν θετική για τη συνέχιση δεν ήταν εις βάρος του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Κυρία Μονίθ, έχει το λόγο. Παρακαλώ σύντομα, σύντομα, σύντομα, ναι, σύντομα πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για κάτι το σημαντικό που είναι αυτοκινοδρόμος της Καντάβριας. Εδώ ήδη η χάραξη αρχική άλλαξε και από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση και δεν ήταν η πρώτη χάραξη από το ΕΛΚ. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε παρόμοιες συζητήσει. Άλλαξε όμως η κυβέρνηση, η σοσιαλιστική αυτή τη χάραξη του δρόμου που ε, πάντα ανησυχούμε, θέλουμε να σεβαστούμε το περιβάλλον και να είμαστε νόμιμοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και ισπανικά πρότυπα και όλα αυτά άλλαξαν λοιπόν και όλα αυτά τα παράπονα που ακούστηκαν ε, ε όπως είπε και ο εκπρόσωπος Επιτροπής, όλα αυτά έκλεισαν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είδαν, πιστοποίησαν, διαπίστωσαν ότι δεν παραβιαζόταν καμία οδηγία για το περιβάλλον, οτιδήποτε πολιτιστικά αν θέλουμε, δικαίωμα και άλλα παρόμοια. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος ε, παρά να κλείσει το θέμα αυτό και μάλιστα για τρίτη φορά, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παλιά και ταπεινά ταπεινά εγώ είπα πέρα από το ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά όλε αυτέ οι αναφορέ όπου διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε, καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, αυτέ θα πρέπει να κλείνουν άμεσα σαν θέμα και έτσι να αποφύγουμε τώρα αυτέ οι συζητήσει ε, και σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών προσφύγοντα σε εμά. Βέβαια θα πρέπει να δούμε τι γίνεται να μην είναι μέσω πολιτικής αναταραχής, μέσω και των μέσων ενημέρωση, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να τους πούμε ότι πρόκειται α πούμε για το 85-337 διάφορα τεχνικά περίπλοκα θέματα. Το αποτέλεσμα όμω το πόρισμα είναι απλό. Όλοι αυτοί που έχουν να κάνουν με το αν σε αυτό το επίπεδο το νομικό εάν υπήρξε μια ε, παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, όλοι αυτοί ε, είπαν ότι δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να το λέμε ότι από τη στιγμή που γίνεται κάτι τέτοιο δεν υπάρχει καμία διαπίση παραβίαση, θα πρέπει να κλείνει η υπόθεση. Κύριε Γκουτιέρες. Εγώ ξέρω τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Χάλασε η η εικόνα η όλη. Όπως ε, ελέγχθη πρέπει να σας πω ότι είναι οι περιοχές αυτές αγροτικές και απ' την άλλη πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία προσφυγή κατά των Ισπανικών αρχών. Επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε μία παράξενη κατάσταση. Βρισκόμαστε στην εξή κατάσταση. Ποτέ όταν ε, εφαρμόζεται η οδηγία περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν γίνεται λόγος για προστασία της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεδομένου ότι όταν καταστραφεί το περιβάλλον δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρατηρήσεις που γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πω ότι συμφώνησαν οι πάντες για να γίνει αυτή η καταστροφή. Κυρία Μουνιές, μου φαίνεται ότι οι αντιφάσεις εδώ είναι τρομερές. Δεν μπορεί κανείς να θέλει για την ε, μόρφια να λέμε ότι εφόσον έχουν γίνει σωστά τα πράγματα, αρχιοθετείται η υπόθεση και τελείωσε και εδώ για αυτή την ε, ε, συγκεκριμένη ε, καταγγελία, για αυτή την αναφορά, παρά το γεγονός ότι τα πάντα έχουν γίνει νομότυπα, να θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Κυρία Γκουτιέρεθ, πρέπει να σας πω ότι η δικαστική οδός και η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή που ακολουθούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στα εθνικά δικαιοδοτικά τους όργανα Εάν όμως εμείς αρχιοδετήσουμε μία υπόθεση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν οι πολίτες να προσφύγουν στα δικά τους δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο λέμε εδώ. Η Επιτροπή Αναφορών ε, πρέπει να αποφανθεί εάν όντω υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Και όπω λένε οι εμπειρογνώμονε και οι υπεύθυνοι τώρα σε σε όλη κατάσταση, καθώ και οι Κομισιόν, Εφόσον μας ότι δεν υπάρχει τέτοιου παραβίαση, το λογικό θα ήταν να αρχιοθετηθεί αυτή η αναφορά που έχει στην περίπτωση της Μούρθια ή όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως, όπως λέω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτε στα εθνικά δικαιοδοτικά του όργανα. Νομίζω ότι ο πρόεδρο ήταν απόλυτα σαφή η ενημέρωση τη Επιτροπή. Δηλαδή, δεν βλέπει να υπάρχει παραβίαση. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να κλείσουμε την υπόθεση. Κυρία Γκουτιέρεθ, εσείς αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας προσφέρετε νέα στοιχεία για την υπόθεση αυτή, λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι κλείνει αυτή η αναφορά, μπορείτε. Βάλτε, ακούστε. Η καταστροφή στο περιβάλλον είναι δρόμος χωρίς γυρισμός. Εάν ένας η ε, ρηπανθεί όπως γίνεται στην Ισπανία, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, τι γίνεται. Γίνεται ένα κακό το γίνουμε να γίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αν ναι, εγώ μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει καταστροφή ολοκληρωτική, δεν μπορούν να συνεχιστούν τα έργα. Τώρα, είναι κάτι το διαφορετικό αν κάποιος έχει δικαίωμα να ρηπαίνει έναν ποταμό ή όχι. Η οδηγία για τις επιπτώσεις των περιβαλλον... για τις αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μένα καπελώνει όλα τα άλλα. Αυτή θα πρέπει να εμφανιστεί. Τώρα, στις ε, περιοχή αυτή, αυτά τα σπήλαια στο παρελθόν, ζούσαν πάρα πολλά άτομα και έχουμε πάρα πολλά σπήλαια, δεν έχουμε ένα, αλλά πρέπει να τα διασώσουμε. Κυρία Γκουτιέρετ. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα προηγουμένω. Αυτή η αναφορά κλείνει. Παρόλα αυτά, μετά από αυτά τα οποία είπατε, εάν θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτό το θέμα με επιχειρήματα. Σε μια άλλη αναφορά μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ λέω να μην κλείσει. Εγώ λέω να μην κλείσει. Δεν λέω να κλείσει. Διότι καταστρέφονται εδώ η, τα σπήλαια. Και το θέμα της ε, καταστροφής χωρίς ε, του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να υπερισχύσει αυτό το επιχείρημα. ο κανόνας είναι ότι όταν ένας βουλευτής ή μία βουλευτή ζητά να παραμείνει ανοιχτή μία υπόθεση, θα πρέπει να την ακούσουμε. Αν θέλει η κυρία Γκουτιέρε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τα σημεία 13 και 14 θα τα συζητήσουμε την επόμενη συνεδρία όχι σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, πέντε λεφτά διάλειμμα και μετά αρχίζει η συνεδρία των συντονιστών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ.